Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Συνεχίζουμε τις χθεσινές μας συνομιλίες. Σημείο 46, προετοιμασία, η συζήτηση μάλλον του σχεδίου εκθέσεως του κυρίου Τσέλερ για την Επιτροπή, εκτέλεση του προϋπολογισμού της Επιτροπής και τον λοιπόν. Ο κύριος Σέλλαρ θα ξεκινήσει. Την παρουσία και του Επιτρόπου Ετιγκερ, ο οποίο είναι και παρόν, τον καλωσορίζω. Κύριε Τσέλλαρ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να πάμε. γρήγορα, γρήγορα. Λοιπόν, έχουμε το σχέδιο της εκθέσεώς μας, της εκθέσεώς μου, αρκετά ογκώδης έκθεση. Θα επικεντρωθώ όμως στην παρουσίαση στα πιο ουσιαστικά. Γιατί είχαμε ούτως άλλως μια δυνατότητα από το Σεπτέμβριο που έχει ξεκινήσει αυτή η συνεδρίαση και με την ακρόαση με τους γενικούς διευθυντές και με τους επιτρόπους, αλλά ιδιαίτερα τον Επίτροπο Έτιγκερ, να συζητήσουμε τα επιμέρους ζητήματα. Απαλλαγή λοιπόν 2016 για την Επιτροπή. Δεν ξέρω αν τα θυμάστε. Τώρα που έχουμε φτάσει στο 16, στο 18. Είχαμε συζητήσει τότε με την έκθεση ότι θα ήταν σκόπιμο να επιταχύνουμε τις διαδικασίες της εκτέλεσης για να είναι πιο κοντά στο έτος για το οποίο δίδεται η απαλλαγή. Για να δούμε αν θα τα καταφέρουμε και ιδιαίτερως θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο, τον Κλάους Χαϊνελένε, τον Πρόεδρό του, τον κύριο Λάζαρο Λαζάρο, τον Αντιπρόεδρο, αλλά και τους λοιπούς συναδέλφους του Ελεκτικού Συνεδρίου για τις ε, πυκνές επαφές και στη συνεργασία. Επίσης θέλω να ευχαριστώ τον Επίτροπο, αλλά και όλους ιδιαίτερους εκείνους που είχαν να ανασκώσουν το μεγάλο βάρος της απαλλαγής έλας και Γκότς της γραμματείας της Επιτροπής Απαλλαγής. Τον κύριο Σέχη από την ε, ομάδα μας και τον Λουκάς Ράιχελ, από δική, ε, το δικό μου βοηθό, χωρίς τον οποίο δεν θα μπορέσει να κάνω αυτή τη δουλειά. Αυτά λοιπόν για τα προκαταρκτικά. Τώρα για το 2016 συγκεκριμένα και την εκτέλεση του προπολογισμού. Τι πρέπει να κοιτάξουμε ιδιαίτερος. οι προτάσεις μας και οι συστάσεις μας έχουν τελικά ενσωματωθεί όπως ε, άλλωστε θα έπρεπε και στους ε, στόχους Επιτροπής και Κοινοβούλιο όπως τους είχαμε ορίσει γιατί είχαμε πολλές προτεραιότητες που πήγαν από τα 10 στα 7 στα 5 χρόνια σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία πολλά αλλάζουν, πολλές προτεραιότητες μετατοπίζονται. Αλλά βέβαια και αντίστοιχε εντολέ και η πολιτική έμφαση που δίνεται σε διάφορα ζητήματα. Επομένω, θα ήταν καλό να έχουμε αυτή την ε, ορατότητα. Επίση, στην αξιολόγηση. Με την επισκόπηση που θέλουμε να κάνουμε, θα ήταν καλό να έχουμε μια εικόνα γενικότερη της χρονικής περίοδου στην οποία αναφερόμαστε και για τις επιμέρους πολιτικές πρέπει να συζητήσουμε τα νέα στοιχεία στην γεωργική πολιτική όπως είναι το πρασίνισμα, το greening, αλλά και ιδιαίτερα προγράμματα όπως ε, αυτό της ενίσχυσης των νέων γεωργών για να αξιολογήσουμε την αποδοτικότητά του και αντίστοιχα. Αλλά, επίσης, η συμπληρωματική υλοποίηση των προγραμμάτων από την πολιτική συνοχής με την ταχύτερη, όπως έχουμε ζητήσει, ε, εκτέλεση των πληρωμών και την αναφορά στον νησιν 2. Είναι κάτι το οποίο είχαμε δει στην προηγούμενη περίοδο προγραμματική περίοδο. Και μετά έχουμε και τον κανόνα να συν 4. Οπότε πρέπει να δούμε τι σημαίνει ή τι συμβαίνει καλύτερα όταν έχουμε ουσιαστικά πολύ μεγάλες καθυστερήσεις και αντίστοιχα βέβαια προβληματική απορρόφηση των ε, πόρων με τον ίση 4. Ίσως θα πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας για την επόμενη προγραμματική περίοδο, έτσι ώστε αυτές οι αποκλήσεις μεταξύ της νέας περίοδου, της νέας προγραμματικής περίοδου και της προηγούμενης να ε, μείνουν σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Επίσης το Κοινοβούλιο ζητεί η Γενική Διεύθυνση να διατυπώνει σε δημόσιο έγγραφο τις συστάσεις της για το κάθε κράτος. Εμένουμε ε, σε αυτό στη διαφάνεια για τη χρηματοδότηση της ε, πολιτικής για, τη μετανα... για το μεταναστευτικό. Έχουμε μια νέα πρόκληση στο πλαίσιο του πολιτού δημοσιονομικού προγράμματος να αντιμετωπίσουμε και πιστεύουμε ότι πρέπει να βελτιωθεί η διαφάνεια και τη γνωρίζουμε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε μια νέα πρόκληση η οποία πιέζει και χρονικά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως, χρειάζονται μέθοδοι και διαδικασίες που θα μας εξασφαλίσουν μια καλύτερη ή ταχύτερη αντίδραση σε αυτές τις προκλήσεις. Και διατυπώνουμε στην ε, έκθεση 2016, διατυπώνεται στην έκθεση 2016 από την Επιτροπή η σχετική πρόθεση που υποστηρίζουμε και εμείς για δε τη μελλοντική ε, περίοδο για το μελλοντικό δημοσιονομικό προγραμματισμό. Πρέπει να προβλεφθεί ειδική γραμμή και προσέγγιση στον προϋπολογισμό. με ανάκτηση κονδυλίων από άλλες γραμμές. Επίσης, το θέμα της διοίκησης και γενικότερα των τελών, της διαχείρισης και των τελών των ε, δημοσιονομικών μέσων, ε, παραδείγματι για την ΕΤΕΠ, τα καταποκοπήν ποσά. Βλέπουμε ότι είναι πολύ υψηλά, όπως το βλέπονται, γιατί αρχικά είχαν προβλεφθεί τα κονδύλια, τα ποσά αυτά για άλλους στόχους και όχι για τη διαχείριση οργανώσεων, εταίρων που καλούνται να υλοποιήσουν τα προγράμματα. Επίσης, όπως είχαμε πει εξ αρχής, επιτάχυνση της διαδικασίας για την απαλλαγή μέσα σε ένα χρονικό πλαίσιο του νη ένα, θα ήταν ευκταίο. Είναι μια πρόκληση την οποία πρέπει να ε, επιδιώξουμε να υλοποιήσουμε. Και κάτι ακόμη, πέραν των προκαταβολικών όλων αυτών, θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όλους τους φίλους και συναδέλφους, τους και ηγητές που συνέβαλαν στην διαβούλευση. Χαίρομαι για τη συζήτηση και βεβαίως προσβλέπω στη συνεργασία για να διατυπώσουμε το υλικό κείμενο της έκθεσης. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Να δώσω τον λόγο στους κοιόδης εισηγητές, σε όσους είναι παρόντες. Κύριε Λαμπάγιοβα, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επιτροπέ, συνάδελφοι. Πρώτα απ' όλα οφείλω να επενέσω τον κύριο Τσέλερ για το πάρα πολύ καλό σχέδιο έκθεσης του γιατί αποτελεί μια πολύ καλή βάση για τους κοιόδης εισηγητές και για όλα τα μέλη της Επιτροπής μας. Εκτιμώ ιδιαίτερο το κεφάλαιο για τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού της κοινότητας, καθώς περιέχει πολλά πράγματα τα οποία είχα θίξει όταν ξεκινήσαμε την απαλλαγή του 16 το προηγούμενο φθινόπωρο. Θα ήθελα έτσι να τονίσω την ε, σημασία της ποιότητας των δεδομένων της απόδοσης, ε, η λεγόμενη δήλωση διαβεβαίωσης ε, για την απόδοση και θα ήθελα άρα να ρωτήσω τον κύριο Επίτροπο καθώς η σημασία αυτών των δεδομένων είναι πάρα πολύ σημαντική, η ποιότητα αυτών των δεδομένων είναι πάρα πολύ σημαντική, ε, ποιε είναι οι δεσμεύσει τη Κομισιόν για την βελτίωση της ποιότητας. Τέλος, ε, θα ήθελα να πω ότι χάρηκα που άκουσα αυτή την εβδομάδα ότι πρέπει να τονιστεί η ενότητα του κοινοτικού προπολογισμού για να προωθήσουμε κάποιες εξελέξεις που δεν μπορούν να επιφέρουν τα κράτη-μέλη μόνα τους και τέλος ε, να έχουμε κάποια προοπτική από τις εισφορές των κρατών μελών στην ε, προστιθέμενη αξία της Ένωσης και νομίζω τα είπατε αυτά και εσείς ε, κύριε Επιτροπέ και θεωρώ επίσης ότι θα πρέπει ο προπολισμός να παρουσιάζεται με βάση τους πολιτικούς στόχους του ΠΔΠ και όχι μόνο αν τομέα. Και το ερώτημά μου είναι το εξή. Ε, και νομίζω ότι θα μπορούσε να μας πει κάτι και ο κύριος Επιτρόπος. Τι διδάγματα άντλησε η Κομισιόν να το τρέχον πιδελταπή για να μην επαναλάβει τα ίδια λάθη το επόμενο. Ποιες είναι οι προθέσεις της Κομισιόν για να αλλάξει την εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Βρυξελών, όπως λέμε, στα μάτια των πολιτών, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το πιο δύσκολο καθήκον που έχουμε τους επόμενους μήνες. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ και σας ε, κύριε Τσέλερ. Ο κύριος Τάραντ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βεβαίως ο εισηγητής να έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά όσον αφορά την απαλλαγή των δαπανών της Κομισιόν και βεβαίω ε, πρέπει να τονίσουμε κατά την απόψή μου ότι η έκθεση παρουσιάζει ξεκαθαρά την διαφορά μεταξύ του εκτιμόμενου ποσοστού σφάλματος που παρουσιάζει το ελεγκτικό συνέδριο και η Κομισιόν, και κατά την προσωπική μου άποψη το ποσοστό αυτό, η μέθοδος ε, αυτή δεν είναι η καλύτερη γιατί τότε έχουν ε, ξοδευτεί τα χρήματα ήδη. αλλά πρέπει να το δούμε αυτό το πώς δηλαδή ξοδεύονται τα ευρωπαϊκά κονδύλια για να βελτιωθεί η κατάσταση στο μέλλον. Το δεύτερο. Η έκθεση βλέπει επικριτικά το ότι υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στις ε, πληρωμές ε, και μπορούμε να το περιγράψουμε ως ένα είδος ε, χρέους του κοινοτικού προϋπολογισμού και επίσης ασκεί κριτική στην αυξημένη χρήση ε, χρηματοπιστωτικών μέσων και εδώ πέρα ο συγητής δικαίως ζητάει να υπάρξει αυξημένος έλεγχος αυτών των μεθόδων. Τέλος. Είναι ίσως μικρά τα ποσά και ίσως δεν αξίζει να το αναφέρουμε αλλά η παράταση της ε, περίοδου αδράνειας θα έπρεπε νομίζω να αφορά και τα μέλη της ε, Κομισιόν και η άποψη της Επιτροπής ε, Δεοντολογίας θα πρέπει να δημοσιεύεται γιατί όταν μιλάμε για ειδικού συμβούλους των επιτρόπων βλέπουμε κάποιους πρώην επιτρόπους εκεί. και οι νυν επίτροποι έχουν μεγάλη διακριτική ευχέρεια στις προσλήψεις αυτών των ειδικών συμβούλων που δουλεύουν όμως ε, με μερική απασχόληση και άρα ταυτόχρονα έχουν άλλα συμφέροντα στον ιδιωτικό τομέα. Οπότε πέρα από την αμοιβή τους, από την Κομισιόν, πρέπει να εξετάσουμε και ε, πιθανή σύγκρουση συμφερόντων και δεν θα πρέπει να περιοριστούν οι έλεγχοι μόνο στο χαρτοφυλάκιο του Επιτρόπου που συμβουλεύουν, καθώς έχουν ανεμπόδιστη πρόσβαση σε ολόκληρη την Κομισιόν, ενώ διατηρούν θέσεις στον ιδιωτικό τομέα. Εγώ δεν μπορώ να μπω, παραδείγματος χάρη, τόσο εύκολα στα κτίρια της Κομισιόν, αλλά με το σήμα του Ειδικού Συμβούλου ε, υπάρχει κανένα πρόβλημα, μπαινοβγαίνεις παντού και Δεν είναι νομίζω σωστός τρόπος αυτός αντιμετώπισης. Του των λεχθέντων θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω τον εισηγητή και την Κομισιόν γιατί τα περισσότερα λεφτά έχουν διατεθεί σωστά. Έχω δύο συναδέλφους ακόμα στον κατάλογο. Ο κύριος Πυρίνσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον ε, κύριο Ζέλερ για την ε, πολύ σωστή και σε βάθος αντιμετώπιση του θέματος. Πιστεύω ότι είναι δικαιολογημένα τα σχόλια ε, και είναι αιτιολογημένη και η σε βάθος ανάλυση αυτή του έτους 2016 γιατί ε, πρέπει να δούμε ποια είναι τα διδάγματα τα οποία μπορούμε ε, να αποκομίσουμε από την εμπειρία. Επίσης συμμερίζομαι την εστίαση που έκανε στην παρουσίασή του στο θέμα των κονδυλίων από το Ταμείο Συνοχής Επίσης, το γεγονός ότι υπογράμμισε τις καθυστερήσεις που έχουν ε, καταχωριστεί το, ε, τον κίνδυνο συσσόρευσης των καθυστερήσεων με αποτέλεσμα στο τέλος της προγραμματικής περίοδου ε, να εκκρεμούν ακόμα πολλά κονδύλια πληρωμών. Πιστεύω ότι αυτά είναι πολύ σοβαρά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να λυθούν γιατί τώρα μπαίνουμε στην ενεργή περίοδο για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Ήδη δουλεύει το προσωπικό και οι αρμόδιοι για τον καθορισμό του, ε, της νέας προγραμματικής ε, περίοδου και επομένως τίθενται ερωτήματα. Μπαίνουμε σε αυτήν τη νέα περίοδο και η Κομισιόν αποφάσισε και λέει ότι θέλει να διασφαλίσει ότι τα προγράμματα θα είναι υψηλής ποιότητας, υψηλής ποιότητας εταιρικές συμφωνίες και επομένως πρέπει να μελετηθούν σωστά τα προσχέδια εταιρικών σχέδιων, σχεδίων να ξανασταλούν προς διόρθωση στις ε, ε, χώρες να ε, μελετηθεί το κατά πόσο αν υπάρχει η εξάντε ερεσιμότητα κλπ. Αυτό θα πρέπει, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί έτσι ώστε να βρούμε τη σωστή ισορροπία ανάμεσα σε δύο πράγματα. Αφενός την εξάντε ε, ε, διαδικασία έτσι ώστε δηλαδή όντως τα προγράμματα είναι σωστά και αφετέρου να, να ε, δαπανηθούν τα χρήματα εν ευθέτω χρόνο. Κυρία Πρόεδρε, πιστεύω ότι θα πρέπει να δούμε το θέμα αυτό και από την πλευρά των μεγάλων προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε όσον αφορά το ευρωπαϊκό πρόγραμμα που είναι η έλλειψη ε, ε, ε, συγγνώμη, οι ανισότητες. Αυτές οι ανισότητες που μπορεί να είναι κοινωνικές φυσικά, αλλά μπορεί να είναι και εδαφικές και άλλες. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στην εξέφραση της σωστής ισορροπίας. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ε, στην προγραμματική περίοδο, όταν προγραμματίζουμε δηλαδή, όταν επικυρώνουμε και ε, θα πρέπει οι διαδικασίες να προχωρούν όσο γίνεται πιο γρήγορα. Βασικά υπάρχουν δύο δυνατότητες. Μπορεί κανείς να είναι πολύ προσεκτικό στην αρχή, να διασφαλίσει τα πάντα και μετά να ξεκινήσεις, αλλά υπάρχει και μία άλλη προσέγγιση, η οποία συνίσταται ε, στο να είναι κανείς όσο γίνεται πιο προσεκτικός, αλλά εν πάση περιπτώσει να προχωρήσει γρήγορα στην πρώτη ε, φάση και μετά να είναι πάρα πολύ αυστηρός και να επιβάλλει πολύ αυστηρές κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων πιστεύω ότι θα πρέπει να συζητήσει και να μελετήσει τα θέματα αυτά η Κομισιόν. Στην έκθεσή σας, κύριε συνάδελφοι, έχετε μία ε, ε, ε, γενικά θετική θεώρηση της εξάντε διαδικασίας. Αναρωτιέμαι εάν απλώς θα πρέπει να εγκρίνουμε ας πούμε αυτή την πρακτική ή μήπως θα πρέπει να δούμε εάν αυτή η εξάντε διαδικασία είναι η εξαντια διαδικασια ειναι ιδέα. Καλωσορίζω λοιπόν και καλοδέχομαι αυτήν την ευκαιρία που έχουμε τον Επίτροπο Έτιγκερ μαζί μας και ευελπιστώ ότι πραγματικά θα θίξει και το θέμα αυτό και θα είναι ένα θέμα για το οποίο θα ακούσουμε ε, κάποια στοιχεία στη διάρκεια αυτής ε, της διαδικασίας απαλλαγής μας απασχολεί σήμερα το πρωί. Ευχαριστώ θα μιλήσω κι εγώ. Θα ήθελα να πω ότι με ευγνώμων για το ότι καλύπτει πλήρως την δουλειά μας η έκθεση αυτή, όλα όσα μας απασχόλησαν και τις αποστολές που κάναμε σε Ουγγαρία και Πολωνία και η Ελλάδα επίσης περιέχεται και επί τη ευκαιρία θα ήθελα να πω δύο λόγια για την Ελλάδα. Είχαμε πάει την προηγούμενη εβδομάδα και αυτό το οποίο είδαμε με τα 181 έργα προτεραιότητας από τα διαρθρωτικά ταμεία είναι οπωσδήποτε μεγάλη επιτυχία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν τίθεται ζήτημα. Είδαμε πάρα πολλά καλά έργα τα οποία οπωσδήποτε θα βοηθήσουν την Ελλάδα και χαιρόμαστε γι' αυτό. Εδώ και χρόνια ασχολούμαστε με το κτηματολόγιο και νομίζω ότι πρέπει να προσέξουμε οι τελευταίες οργανωτικές αλλαγές να μην καθυστερήσουν την ε, κατάσταση γιατί πρέπει να υποβάλουν ε, όλοι οι εργαζόμενοι ξανά αίτηση για την θέση τους ε, από ό,τι φαίνεται οπότε πρέπει να μεταδώσουμε σε όλους το μήνυμα ότι πρόκειται για ένα, κλειδί, για ένα έργο κλειδί και για την Ελλάδα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και χρειάζεται να ολοκληρωθεί νομίζω το 2020 και συνολικά θα έλεγα ότι είχαμε μια πάρα πολύ καλή εντύπωση, πολύ καλοί διαχειριστές ε, κάνουν καλά τη δουλειά τους και όπου υπάρχουν στεποί στην εφαρμογή των αποφάσεων παραδείγματος χάρη όσον αφορά τις απαλωτριώσεις και αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να λυθούν με την βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καλό θα ήταν νομίζω ακριβώς αυτή τη μεγάλη επιτυχία να τη μεταδώσουμε και προς τα έξω. Δεύτερον, συνάδελφος ο κύριος Τσέλερ σωστά επισημαίνει ότι πρέπει να γίνει πιο σύντομη η διαδικασία της απαλλαγής πρέπει η όλη διαδικασία να ολοκληρώνεται σε ένα χρόνο νη ένα. Δηλαδή να σκεφτούμε ότι ε, οι εταιρείε ε, κάνουν μέσα σε τρεις μήνες ε, τον ισολογισμό τους και εμείς ένα χρόνο και ένα μισή θα πρέπει να γίνουμε κάπως καλύτερη και πρέπει ακριβώς να τα καταφέρουμε. Έχω μία ερώτηση ε, σε ένα μέρος ε, του σχεδίου έκθεσης. Ε, αυτό το οποίο αφορά το πρασίνισμα και τους νέους αγρότες. Το ερώτημα είναι και το ελεγκτικό συνέδριο αποκάλυψε ότι υπάρχει μεγάλη λανθασμένη χρήση των ε, κονδυλίων. Ε, δεν είναι απλό, αλλά δεν μπορεί να αφήσουμε να συνεχίζεται έτσι αυτή η υπόθεση. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε το τι μπορεί να γίνει σε αυτά τα θέματα, γιατί μιλάμε για σημαντικά κονδύλια και βεβαίως ε, υποθέτουμε ότι θα πρέπει να δούμε το τι θα γίνει με την επιστολή που είχαμε απευθύνει με τον κύριο Τσέλερ για προς την ε, Κομισιόν για τις συστάσεις που είχαμε κάνει. Κύριε Επίτροπε, έχετε τον λόγο. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ καταρχάς για τη συνεργασία με τους επιτρόπους. Εν προκειμένου, στη συνεργασία σας, στη διαδικασία αυτή για την απαλλαγή, πιστεύω ότι ο κύριος Τσέλερ και οι οι συναδελφοί του έχουν διατυπώσει πολύ θετικέ συστάσεις. Το να έρθει πιο νωρίς λοιπόν, να ολοκληρωθεί ταχύτερα, να εντατικοποιηθεί ε, και να γίνει πιο απρόσκοπτη αυτή η διαδικασία της απαλλαγής θα είναι ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα. Εσείς από εμά περιμένετε δηλαδή να ε, επιταχύνουμε τη διαδικασία να την εντατικοποιήσουμε. Και βεβαίω αυτό αφορά και τους συναδέλφου μου και τις υπηρεσίε μου και εμένα προσωπικά. Σαν έτοιμα. Έχω το ίδιο θέμα να συζητήσω σήμερα το μεσημέρι, απαλλαγή 2016, με το Συμβούλιο. Το Κοινοβούλιο έχει ιδιαίτερη γνώση και εξειδίκευση στο θέμα της απαλλαγής και τον έλεγχο του προπολογισμού. Το Συμβούλιο είναι συμβούλιο το οποίο δεν έχει να ασχοληθεί μόνο με δημοσιονομική πολιτική και πολιτική για την, ε, την απαλλαγή, αλλά νομισματική, οικονομική πολιτική και, και γενικότερα θέματα. Και έτσι η απαλλαγή δεν είναι πάντα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και της δουλειάς του Συμβουλίου όπως είναι τη δουλειά του Κοινοβουλίου. Θέμα προτεραιότητας το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο παραδείγματι του προηγούμενου έτους θα μπορούσαμε να είχαμε ε, φέρει πιο νωρίς τον, ε, το θέμα της απαλλαγής για το 2016. Αλλά ήταν η ώρα να συζητήσουμε τον προπολογισμό ε, του 2019. Ή η χθεσινή συζήτηση που είχαμε την επιλογή του Αντιπροέδρου του της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Επομένως, αυτό εξαρτάται πάντα η επιτάχυνση των εργασιών από τον Προεδρεύοντα και τη Γραμματεία του Συμβουλίου. Εκείνοι προσδιορίζουν με όλη την ε, θεματολογία και την επιβάρυνση του ημερήσιας διάταξης που έχουν στο Συμβούλιο ποιο θέμα θα φέρουν πιο μπροστά. Όπως είπα, η απαλλαγή θα μπορούσε και πέρσι ακόμα για το προηγούμενο έτος να είχε κλείσει. Να μην περάσει στο δεύτερο έτος, στον 2. ομολογώ ότι και εγώ πολλέ φορέ μπερδεύομαι. Πρέπει κάθε φορά να κοιτάω. Για ποιο συζητάμε τώρα, 14, το 15, το 16, ποια από όλα τα έτη έχουμε. Ε, μην ξεχνάμε όμω ότι έχουμε και τι εθνικέ ε, διαδικασίε για την απαλλαγή από τι οποίε εμεί είμαστε συνηθισμένοι, γιατί είναι ε, πιο γρήγορε. Και επίσης, το πλαίσιο αυτό, το δημοσιονομικό, 21, 27. Δεν έχουμε προχωρήσει. Έχουμε εκλογές το 19. Θα ξαναεκλεγούν οι βουλευτές. Μετά θα έχουμε την Επιτροπή. Αλλά η χειρότερη περίπτωση ποια θα ήταν, το worst case scenario. Νέα Επιτροπή το, το Νοέμβριο του 2019 να αναλάβει καθήκοντα με 27 επιτρόπους, να αρχίσει να ασχολείται με ένα δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο ποτέ θα είναι έτοιμο. Δεν θα είναι έτοιμο δηλαδή πριν το 2020, δεν θα είναι έτοιμο εγκαίρως. Και άρα μόνο το 2022 θα έχουμε το νέο πλαίσιο. Σκεφτείτε τώρα τον, ε, τη διαδικασία όλη που προβλέπει τη συμμετοχή των ε, εθνικών, τοπικών, περιφερειακών αρχών, κυβερνήσεων κτλ. Οι δε εταίροι μας, όλοι όσοι έχουν να κάνουν τον προπολογισμό, περιμένουν από εμά, περιμένουν από το Κοινοβούλιο, να ετοιμάσει εγκαίρω και μαζί με το Συμβούλιο το πολιτεύσιο δημοσιονομικό πλαίσιο. Υπάρχει άτυπη συνάντηση των 27 αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων αυτή τη βδομάδα για να προσδιορίσει και θα έχει τεράστια σημασία τις ε, κατευθύνσεις και το εάν είναι διατεθειμένοι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων να ορίσουν ως προτεραιότητα το σχεδιασμό του πολιτούς δημοσιονομικού πλαίσιου και να το κλείσουμε στο 18. Και σας λέω πολύ συγκεκριμένα πώς θα ξεφύγουμε από το ε, περιορισμό του 1,0 στην αύξηση του προπολογισμού, του πολιτικού δημοσιονομικού πλησίου. Είναι πραγματικά πολύ στενά αυτά τα περιθώρια. Πρέπει να βρούμε λύσεις. Μην ξεχνάμε ότι κι εσείς από εθνικούς εκλογικούς ε, καταλόγους υποψηφίων προέρχεστε, δεν υπάρχει ευρωπαϊκή, ε, ευρωπαϊκό δηλαδή, ευρωπαϊκή εκλογική λίστα, ευρωπαϊκός κατάλογος υποψηφίων. Και άρα είστε κι εσείς σε αυτό περιοριζόμενοι από το 1,0. Εγώ κάνω προβλέψεις με κάτι περισσότερο. Αλλά καθήκον δικό μας, ολονών αλλά και δικό σας. Και το λέω εγώ και για όσους είναι από την Αυστρία, από την Ιρλανδία, από τη Σουηδία, από τη Φιλανδία, τη Δανία, από τη Γερμανία, να καταστήσετε σαφές και στα κράτη-μέλη ότι με αυτό το στενό κορσέ του 1,0 συνοχή, μετανάστευση, γεωργία, άμυνα δεν θα βρουν αντάξια ανταπόκριση και λύσεις. Αυτό θέλω να το πούμε ξεκάθαρα. Και έχουμε ένα εφταετές πολιτές στο πλαίσιο επτά ετές για τελευταία φορά προτείνεται. Θα ήμουν ευγνώμων η κυρία Τομά και ο κύριος Σούλμπριχτ, οι δύο εισηγητές σας, να κάνουν τη δουλειά με αυτή την προοπτική ακριβώς του επταετούς δημοσιονομικού πλαισίου που προτείνει η Επιτροπή, αυτή τη στιγμή εμείς δηλαδή, και το οποίο ε, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει να έχουν κλείσει πριν μπουν στην προεκλογική διαδικασία. Με κάθε καλή διάθεση και βούληση νομίζω ότι θα το λύσουμε αυτό το θέμα, θα μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι και οι πρόεδροι των πολιτικών ομάδων αλλά και ο πρόεδρος Ταγιάννη πρέπει μέσα από αυτό το χρονοδιάγραμμα, όπως άλλωστε έχουν λίγο πολύ προσδιορίσει και νομίζω ότι από το Μάιο και μέχρι το τέλος του 2019 θα μπορούμε να έχουμε προχωρήσει αρκετά και οι επιμέρους επιτροπές να προσδιορίσουν και τους εισηγητέ του. Εμεί από πλευρά μα θα κάνουμε με τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια τη δουλειά μα για να είμαστε σε θέση, εάν στι 2 Μαου έρθει να ψηφιστεί αυτό το θέμα, να, να υποβληθεί το θέμα αυτό του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου, να είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε και να ολοκληρώσουμε πριν από τις θερινές διακοπές του 18. Και μετά. Πέντε χρόνια ή πέντε σε πέντε. Και εδώ, κύριε Τσέλερ, κύριε Σναλφέ, έχουμε να κάνουμε με την σύμπτωση των χρονικών αξώνων, δηλαδή την παράλληλη εξέλιξη με τις εκλογές του 19, με την Επιτροπή πάλι την εγκαθίδρυση της νέας επιτροπής που θα χρειαστεί ένα χρόνο λίγο πολύ για να ετοιμάσει τον νέο προϋπολογισμό, να τον συζητήσει και να τον υποβάλει δηλαδή. Και άρα η νέα Επιτροπή από το 2020 και μετά θα πρέπει να έχει θέση σε αυτό το χρονικό περιθώριο. Δεν είναι δυνατόν να μας πιέζετε και να μας υποχρεώνετε να είμαστε έτοιμοι για να υποβάλουμε προτάσεις τρία χρόνια πριν από τις προσεχείς, από τις επόμενες ε, δημοσιονομικές προοπτικές. Τρία χρόνια μας λέτε. Αυτή είναι μια πίεση απαράδεκτη, δεν το βλέπω πουθενά σε καμιά άλλη εθνική διαδικασία. Επομένως πρέπει να είστε κι εσείς διατεθειμένοι να μας επιτρέψετε, δηλαδή όχι σε εμάς, στους επόμενους ε, ε επιτρόπους, στην επόμενη επιτροπή, να έχουν δύο χρόνια προκαταβολή στην υποβολή των προτάσεων, όχι τρία όπως απαιτείται τώρα, δηλαδή μετά το 2020 να έχουμε από το 25 και μετά να υποβάλουμε προτάσεις, όχι από το 2023. Και έτσι θα έχουμε με πενταετή προοπτική 2026 το Κοινοβούλιο να συζητεί το 28 μέχρι το 2030 και το καθεξής τις προτάσεις. Έτσι γλιτώνουμε και από την πίεση με την έννοια ότι το Κοινοβούλιο το 28 προσδορίζει μόνο του τις εκλογές, το προϋπολογισμό, το, πολιτι, το πλαίσιο. Δεν χρειάζεται δηλαδή να πιέζεται από το δικό του εκλογικό χρονοδιάγραμμα και έτσι μπορούν μέσα σε 1,5 χρόνο η Επιτροπή μαζί με το Κοινοβούλιο να είναι έτοιμη μέσα σε 1,5 χρόνο και να έχουν εγκαίρω τις προτάσεις ώστε και ο ερευνητής, ο Γιώργος η περιφέρεια να έχουν τα στοιχεία στη θέση τους, να μπορούν να σχεδιάσουν το, τα επόμενα βήματα με, τα, με το προσεχές πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Να μην χρειάζεται να περιμένουν για να ορίσουν τις αρχές, τη διαχείριση, την εκτέλεση, γιατί χάνονται χρόνια πολύτιμα για ευρωπαϊκές επενδύσεις. Έχω τώρα ερευνητικές ομάδες, ενώσεις γεωργών, ε, τράπεζες επενδύσεων, υποστήριξη των επενδύσεων, την κεντρική, την ΚΑΕΒΕ και τις ε, περιφερειακές των κρατηδίων. Και μου λένε σας παρακαλούμε δώστε μας εγκαίρως στα στοιχεία για να προετοιμαστούμε για το προσεχές δημοσιονομικό πλαίσιο που ξεκινά το 2021. Έχουμε αρκετό χρόνο. Σας το λέω έτσι με έντονους τόνους γιατί δεν υπάρχει περίπτωση αλλιώς να κάνουμε τη δουλειά μας με παράλληλη εργασία εάν δεν επιταχύνουμε λίγο και εμείς και αν δεν αφήσουμε ένα μεγαλύτερο περιθώριο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πέντε χρόνια δηλαδή διάρκεια και δύο χρόνια νωρίτερα, ώστε να μπορούμε και μέσα σε μισό χρόνο να το κλείνουμε, έτσι ώστε να μπορούμε να δώσουμε και στους εταίρους το χρόνο να προετοιμαστούν. Αναφερθήκατε στη μετανάστευση και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Όντως, η μετανάστευση στο εύρος που διατυπώθηκε, που εκφράστηκε το 2011-2012 δεν είδε ευρωπαϊκή ανταπόκριση. Και είναι το νέο μεγάλο καθήκον της Ευρώπης. Μπαίνει στον προϋπολογισμό, πρικοδοτείται τακτικά. Αυτή τη στιγμή δηλαδή έχουμε μόνο μία αντιμετώπιση των προβλημάτων, μία μετακτόπιση κονδυλίων ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν και πρέπει πλέον να δώσουμε απαντήσεις σαφείς με χρηματοδότηση ρεαλιστική, με απαντήσεις αποτελεσματικές από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, αλλά και με τα ταμεία και καταπιστεύματα και από την ε, διακήρυξη κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που μπορούν να δώσουν τις κατάλληλες απαντήσεις. Εν γέννη είμαστε ευγνώμονες προς το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο, το οποίο για πρώτη φορά δίνει μια επιφύλαξη αξιολόγησης, μια σαφή δηλαδή ε, πρόοδο. Το ποσοστό του σφάλματος από το 3,8% στο 2015 έχει πέσει στο 3,1% για το 2016, δεύτερη και σημαντική πρόοδος για την οποία και ευχαριστώ θερμά τους συνεργάτες τους δικούς μου αλλά και τα κράτη-μέλη στην κοινή διαχείριση. Πρόκειται για μια εξέλιξη την οποία οφείλουμε να αποδώσουμε και στη δική σας επικοδομητική στάση. Παρακολουθείτε δηλαδή στενά τη δική μας την ε, λειτουργία και δράση και μας ε, βοηθάτε να κάνουμε τις ορθωτικές κινήσεις. μας σε μια διαδικασία Μάθηση, το ελεγκτικό συνέδριο, η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού, εμείς και το Συμβούλιο βεβαίω πρέπει να παραμείνουμε στην τήρηση αυτών των αρχών και προϋποθέσεων, μαθαίνοντας και από τα ασφάλματά μας ακόμα και διορθώνοντας την πορεία όπου χρειάζεται. Σας το υπόσχομαι ότι θα συνεχιστεί αυτό. Πάντα έχουμε βέβαια τη διελκυστίνδα μεταξύ single order και απλουστεύση αφενός και ενιαίας αντιμετώπιση αφετέρου. Εάν δηλαδή πρέπει για τον κάθε γεωργό να ε, ορίσω και έναν υπάλληλο της Επιτροπής ο οποίος θα παρακολουθεί το πώς λειτουργεί το πρασίνισμα και έναν αντίστοιχα από το κάθε κράτος μέλος τον οποίο θα παρακολουθεί ένας υπάλληλο της Επιτροπής και έναν της Επιτροπής τον οποίο θα παρακολουθεί ένας του Κοινοβουλίου δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να λύσουμε κανένα πρόβλημα αλλά θα επιβαρύνουμε ιδιαίτερα το συνολικό κόστος. Επομένως πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να βρούμε μια ισορροπία λεπτή βεβαίως μεταξύ των πολύ διεξοδικών ελέγχων αλλά και ταυτόχρονα μιας ισχνής και αποτελεσματικής γραφειοκρατίας και διαδικασίας ελέγχου. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου του, του Λουξεμβούργου, που εσείς τον γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα και πολύ περισσότερο χρόνο, γιατί ήταν και από τα ηγετικά στελέχη εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχει οθετήσει μια διαφορετική φιλοσοφία, μια προσέγγιση διαφορετική με ελέγχους ε, και ε, εντοπισμό των σφαλμάτων ε, και διόρθωσή τους. Μια πολύ καλή φιλοσοφία την οποία εγώ την εκτιμώ. Θα δοκιμαστεί βεβαίως, θα αξιολογηθεί και βεβαίως θα υποστηριχθεί. Βεβαίως, καλούμαστε πάντα να εξηγήσουμε ποιο είναι το μέλλον της Ευρώπης και τι προσέγγιση προβλέπουμε γι' αυτό. Η Λευκή Βίβλος και το έγγραφο αναλογισμού είναι υπό επεξεργασία στην Επιτροπή για να δώσουμε έτσι όθηση σε μια ευρύτερη συζήτηση, ένα ευρύτερο δημόσιο διάλογο. Το προηγούμενο Σεπτέμβριο ο πρόεδρος Γιουνκέρ έδωσε τις προοπτικές και τις κατευθύνσεις της Ευρώπης. Τα επόμενα χρόνια θα πρέπει να, κάνουμε την, να εξασφαλίσουμε την ισορροπία μεταξύ των παραδοσιακών καθηκόντων και των νέων προκλήσεων που έχει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί η συνθήκη ορίζει τη συνοχή και την κοινή γεωργική πολιτική ως υποχρεωτικές δαπάνες και καθήκοντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άρα ως πρωτογενές δίκαιο. Αφενός. Αφετέρου όμως πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι έχουμε νέα καθήκοντα και ευθύνες. Μετανάστευση, έρευνα για την άμυνα, άμυνα, εξωτερική ασφάλεια, καταπολέμηση του ιστρομοκρατίας, προστασία των εξωτερικών συνόρων, τα οποία καλύτερα ή μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να υπηρετήσει και αντίστοιχα να χρηματοδοτήσει. Και εγώ πιστεύω ότι η σύγκρουση μεταξύ συνοχή γεωργική πολιτική αφενό και νέων καθηκόντων αφετέρου είναι μια σύγκρουση που πρέπει να αποφύγουμε και πρέπει να βρούμε τη χρυσή τομή μεταξύ των δύο. Αν με ρωτάτε ποιο είναι το όραμά μου για τα επόμενα δημοσιονομικά έτη, τέσσερις μεγάλους στόχους θα αναφέρω. Guiding principles. Οικονομική ευρωστία πρώτον και ανταγωνιστικότητα. Ο ισχυρός όμως ταυτόχρονα πρέπει να, δείχνει και αλληλεγγύη. Άρα αλληλεγγύη είναι ο δεύτερος κύριος στόχος. Όποιος είναι Όποιο δείχνει αλληλεγγύη πρέπει να δείχνει και τη δυνατότητα να διατηρήσει αυτή του την στάση αυτή του την ευρωστία και την ελληνική άρα αηφορία και τέταρτον εξωτερική πολιτική. Αλληλεγγύη, ασφάλεια δηλαδή και όπως είπα οικονομική ευρωστία, αλληλεγγύη, αηφορία και ασφάλεια είναι οι τέσσερις οδηγοί για τα επόμενα χρόνια, για τα 500 εκατομμύρια των Ευρωπαίων πολιτών. Εσείς όπως και η Επιτροπή Προϋπολογισμού ακριβώς βλέπετε ε, και έχετε ασκήσει κριτική στην αργή εξέλιξη των προγραμμάτων μας, ειδικά στον τομέα της συνοχής. Και το ίδιο κάνω και εγώ και βλέπω τρεις λόγους γι' αυτό. Ένας λόγος, το νησιν 3. Τα κράτη-μέλη δεν βιάζονται. Το 2014, 2015 και 2016 ήθελαν πρώτα απ' όλα να πάρουν κονδύλια του 7 με 13. Μόλις το 2017, όταν εξαντλήθηκε το νη συν 3, ασχολήθηκαν με την απορρόφηση κονδυλίων από το τρέχον πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Κάναμε πολλά. Την ε, απέτηση να οριστούν ε, αρχές ε, για να κινητοποιήσουμε τα κράτη-μέλη έτσι ώστε τέλος 2019, 2020 και 2021 να μην επαναληφθεί το ίδιο φαινόμενο που είχαμε 2013 με 2015 και σας δημιουργήσε προβλήματα, δηλαδή πολλά τιμολόγια και ε, οι πληρωμές μετά να μην γίνονται εγκαίρως. Γι' αυτό για μένα το νησιν 2 είναι προτιμητέο στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο θα προτείνω νησιν 2 και όχι νησιν 3. Η ποιότητα των ε, δεδομένων. Και ε, αυτό ε, είναι ένα σωστό ερώτημα. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι για τον προπολογισμό του 2017 θα υποβάλουμε μια συνολική έκθεση για την προέλευση και την ποιότητα των δεδομένων μας στο Κοινοβούλιο. Και εκεί πέρα θα λέμε ποιε είναι οι πηγές των δεδομένων και πώς αξιολογούμε την ποιότητα των δεδομένων ε, είτε προέρχονται από κράτη-μέλη είτε από περιφέρειες. Θα ήθελα επίσης με κάποια περηφάνεια να υπενθυμίσω ότι υπήρξε πρόσφατα μια έκθεση του ΩΣΑ που μίλησε για εξαιρετική ποιότητα της εκτέλεσης και των δεδομένων του προϋπολογισμού μας. Ο από το Παρίσι εδώ και χρόνια αξιολογεί την εκτέλεση και τον έλεγχο του προϋπολογισμού και την διαδικασία ελέγχου με τα κράτη-μέλη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι άξιο πρόσεκτο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο δικός μας ο προϋπολογισμός τα πήγε καλύτερα από την Γαλλία, τη Γερμανία, από χώρες εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι μέλη του ΩΣΑ. Θα ήθελα λοιπόν κάποια στιγμή ε, να καλέσετε εδώ πέρα και τον Γενικό Γραμματέα του ΩΣΑ για να δείτε ότι εντάξει μπορεί να μην είμαστε ε, πάρα πολύ καλοί αλλά είμαστε σαφώς καλύτεροι από τους ομολογούς μας στον δυτικό κόσμο που λογοδοτούν στα κοινοβούλια. Θα έλεγα ότι κανείς δεν είναι σε καλύτερη θέση από ε, εμάς εδώ και Συμβούλιο και Κομισιόν. Τώρα, για τα τέλη αυτά θα πρέπει να δούμε στο επόμενο ΠΔΠ τι ρόλο παίζει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για εμάς. Γιατί υπάρχουν εδώ πέρα μεγάλες αποκλήσεις ε, απόψεων. Είναι ευρωπαϊκή πρώτα απ' όλα Τράπεζα Επενδύσεων. Δικός μας εταίρος λοιπόν και ακριβώς έχει 28, 27 προσεχώς ε, κράτη-μέλη και εκεί πέρα δραστηριοποιείται Βέβαια και η μετοχή της είναι τα κράτη-μέλη, όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό ε, έχει την ε, σημασία του και πρέπει να το δεχτούμε. Επιπλέον εμείς ως Κομισιόν δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να είμαστε πουθενά μέτοχοι. Πριν από ένα έτος, ε, πριν είχα αποφασίσει υπό την παλιά μου ιδιότητα να δώσω το Euronews 25 εκατομμύρια το χρόνο και είχαμε πει ότι δεν θα πρέπει να είμαστε μέτοχοι και ήταν τελικά απαραίτητοι επενδυτές που ζούσαν στο Κάιρο και στο Λονδίνο. Θα πρέπει ίσως κάποια μελλοντική κομισιόν να σκεφτεί μήπως όπως και εθνικές κυβερνήσεις ε, θα έπρεπε να έχουμε την δυνατότητα εκεί όπου έχουμε συμφέροντα να είμαστε και μέτοχοι, όπως κάνει το γαλλικό ή το γερμανικό κράτος με τους σιδηρόδρομους παραδείγματο χάρη κτλ. Γιατί αλλιώς είμαστε αδύναμοι και απλά δίνουμε λεφτά. Το 6% δεν είναι ε, τελείως λάθος. Επίσης στον τίτλο 5 ε, όπου χρηματοδοτούμε ε, προσωπικό και κτίρια υπάρχει και εκεί πέρα πλαφόν 6%. Παρ' όλα αυτά μπορούμε να εξετάσουμε παρά το ότι αλλού είναι μεγαλύτερο το ποσοστό είναι το σωστό ποσοστό με πολύ βεβαίως χαμηλούς κινδύνους για να δούμε αν καλύπτεται έτσι το κόστος και έρχομαι και σε ένα άλλο πιο συναρπαστικό θέμα χαμένες επιδοτήσεις, δάνεια και καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα θα πρέπει να το συζητήσουμε αυτό το θέμα εις βάθος στο πλαίσιο του πι Ποια έργα ε, χρηματοδοτούνται μόνο με επιδοτήσεις και πού μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε νέα μέσα, δάνεια, εγγυήσεις κτλ. Είτε μόνοι μας, είτε συμπληρωματικά σε πλαίσιο ενός πακέτου να γίνουν έργα. Τώρα που μπορουμε να χρησιμοποιησουμε νεα μεσα δανεια εγγυησει κτλ ειτε μονοι μας ειτε αποκτήσει την εμπειρία με το σχέδιο Γιούνκερ ε, θα πρέπει να γίνει μια διαβούλευση πριν από το επόμενο πι. Μπορώ να σας πω ότι και προηγούμενοι επίτροποι ε, όταν ε, γίνονται σύμβουλοι της Κομισιόν συμμορφώνονται στα όσα προβλέπονται σε ζητήματα δεοντολογίας, συμμόρφωσης και σύγκρουσης συμφερόντων. Και είμαστε, θα έλεγα, σχετικά συγκρατημένοι. Βεβαίως, δεν πρόκειται για μια δουλειά πλήρους απασχόλησης, οπότε δεν μπορούμε να τους απαγορεύσουμε να δραστηριοποιούνται κάπου αλλού παράλληλα. Έχουμε τώρα παρατείνει την φάση αδράνειας, δύο έτη για επιτρόπους, τρία χρόνια για τον πρόεδρο της Επιτροπής. Γνωρίζω ότι ε, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στις ε, εθνικές ε, κυβερνήσεις, ούτε για τους βουλευτές. Τρία χρόνια. Δηλαδή, θα φύγει ο Γιούγκερ και μετά θα γράψει τα απομνημονεύματά του. Γιατί, κοιτάξτε, με αυτήν την έννοια δεν θα βρείτε ποτέ μια 40χρονη γυναίκα η οποία θα δεχτεί να κάνει κάτι τέτοιο και μετά θα της πούμε «Α, όταν τελειώσει η θητεία σου θα πρέπει να κάθεσαι κάποια χρόνια». Πρέπει να είναι και ελκυστική η θέση, ειδικά των επιτρόπων. Αλλιώς θα βρίσκεται μόνο γκριζομάλιδες, 55 ε, θα, που θα κάνουν μια θητεία στην κομψιόν και μετά θα χαλαρώσουν τρία χρόνια πριν ε, βγουν στη σύνταξη. Οπότε ας είμαστε κάπως ε, λογική να δούμε το τι θα δεχόμασταν εμείς, ε, αν θα τα κάναμε εμείς αυτά τα οποία θέλουμε να κάνουν οι άλλοι. Και βεβαίως οποιοδήποτε βουλευτής είναι πάντα καλοδεχούμενο. Ελάτε αύριο το πρωί, πείτε είμαι βουλευτή ε, θα σας ανοίξουμε το, θα απλώσουμε το κόκκινο χαλί. Ε, και εγώ επίσης δεν μπορώ με το μπάτζ μου να μπω τόσο απλά. Πρέπει να δώσω το σηματάκι, ε, ελέγχουν τους συνεργάτες μου, πρέπει να δηλώσουμε ποιοι είναι, μας ελέγχουν τις ε, τσάντες θα ήθελα πράγματι μεταξύ του κτηρίου αυτού και του Μπερλεμό της Κομισιόν να υπάρχει μια αμοιβαία σχέση αν θέλετε να έχουμε όλοι δικαίωμα πρόσβασης και εσείς να έρχεστε και εμείς να μπορούμε να μπαίνουμε εδώ πέρα ελεύθερα και στο Στρασβούργο νομίζω το καλύτερο αυτό θα ήταν για τα θεσμικά μας όργανα. Αυτά για την ώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Ε, χαιρόμαστε όλοι που ε, δείχνετε τέτοιο ενθουσιασμό για να έρχεστε στο κοινοβούλιο σε τακτική βάση. Θα δούμε. Μήπως σας δώσουμε και ένα μπάτζ. Ε, η κυρία Γκρέσλερ έφυγε για λίγο, επομένως εγώ θα την αντικαταστήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Επίτροπε για αυτήν την πολύ συνολική έτσι, καθολική αντιμετώπιση Σα Ευχαριστούμε για τα σχόλια. Έχουμε κάποιο χρόνο. Μπορούμε να ε, πάρουμε κάποιε ερωτήσει. Η κυρία Γιάλα Σέντερ έχει εγγραφεί πρώτη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να ζητήσω συγγνώμη πρώτα απ' όλα από τον ε, ε, Επιτροπό Τιγκέρ γιατί ε, αυτή τη βδομάδα έχουμε ένα, μια δέσμη για τους αυτοκινητοδρόμους και γενικώ δεν ήμουν από την αρχή. Εν πάση περιπτώσει πάντως ήρθα και τα κατάφερα και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί άξιζε τον κόπο που άκουσα αυτά που είπε και πραγματικά ε, αποτελούν τροφή για σκέψη τα όσα μου είπε και βεβαίως εκτιμούμε ιδιαίτερος αυτή τη φρεσκάδα που έφερε ε, η ε, αίσθηση του χιούμορ που έχει γιατί ξέρουμε υπάρχουν πολλές δυσκολίες ε, και νομίζω ότι πρέπει να γελάμε και με τις δυσκολίες μας και καλό είναι γενικά και σε τούτη την Επιτροπή λίγο περισσότερο γέλιο δεν θα έκανε κακό. Ναι, πρέπει να το πούμε και στην κυρία Γκρέσλερ να έχουμε λίγο πιο καλή διάθεση και πιο έτσι ε, παιχνιώδη εν πάση περιπτώσει αντιμετώπιση ορισμένων πραγμάτων. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, συμφωνώ με αυτά που λέγατε προηγουμένως, δηλαδή θα πρέπει όντω και εσείς να βρείτε στο Κοινοβούλιο ε, και να μπορέσουμε ε, να πάμε σε ένα πολιετές ε, κατά το ελάχιστο για, με 1,03 γιατί υπάρχουν όντως προβλήματα. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Πολιτική Πολιτική Συνοχής και αυτά είναι τα βαριά χαρτιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επομένως θα πρέπει για αυτά τα θέματα να βρούμε την καλύτερη δυνατή η ισορροπία. Να βρούμε δηλαδή μια φόρμουλα αλληλεγγύης η οποία όμως να είναι καλά ε, ε, προετοιμασμένη γιατί τα τελευταία χρόνια έχουν συσσωρευτεί κάποια, κάποια προβλήματα τα οποία ε, τελικά βάζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση στην πυρά. Γίνεται ο, ο, ο, τράγος κατά κάποιο τρόπο. και γενικά διαπιστώνουμε μία αυξανόμενη καχυποψία ε, για την λεγόμενη γεωγραφική ανισορροπία. Ε, δηλαδή η κατανομή των κονδυλίων ε, είναι κατά κάποιο τρόπο για πολλούς η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών. Ε, και δεν έχει έννοια να σκεφτόμαστε, να ξανασκεφτόμαστε και να ε, στρέφουν όλοι τα βλέμματά τους στην καμινάδα μας να δούμε αν βγαίνει λευκός ή μαύρος καπνός αλλά θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι ε, ε, παίρνουμε τις πολιτικές αποφάσεις οι οποίες πρέπει να ληφθούν και ότι δεν είμαστε ε, όμοιροι ούτε μπορεί να θεωρηθούν τα κονδύλια των διαφόρων ταμείων ε, επιβράβευση ή αντιθέτως κύρος η τιμωρία κάποιων. Ε, είμαστε Ευρωπαίοι και επομένως εμείς θα πρέπει να ολοκληρώσουμε, να φέρουμε εις πέρας αυτές τις δεσμεύσεις ε, για τις οποίες έχουμε δεσμευτεί. Ε, θα, απ' την άλλη πλευρά βεβαίως είναι γεγονός ότι υπάρχουν ε, δημαγωγικές θέσεις, ε, ακούγονται πολλές λαϊκίστικες φωνές κτλ. Δεν μπορούμε να είμαστε όμοιροι όλων αυτών και το τι κάνει το Συμβούλιο ή αν μαλώνουν μεταξύ τους ή δεν συμφωνούν, στο τέλος τέλος αυτό δεν μας αφορά. Ε, νομίζω ότι μία τέτοια στάση θα ήταν το χειρότερο, που θα μπορούσαμε, το χειρότερο δώρο που θα μπορούσαμε να κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, αν θέλουμε να σκεφτούμε λίγο περισσότερο όχι για να δημοπρατούμε, γιατί αυτό έχει αρνητικό πρόσημο, αλλά εν πάση περιπτώσει να έχουμε μία κατανομή η οποία θα βασίζεται σε, λίγο, σε ένα λίγο διαφορετικό ε, σκεπτικό να υπο... για το ΕΦΣΙ, για διάφορα άλλα ε, ταμεία και προγράμματα. Ε, μία καλύτερη αντιμετώπιση των προγραμμάτων που, έτσι, που αυτά να πρέπει να έχουν και προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία αλλά και να αποφύγουμε και τον σκόπελο των, της κακής γεωγραφικής κατανομής. Ε, όταν, ε, γιατί μπορεί να έχουμε προγράμματα τα οποία έχουν μεγάλη προστιθέμενη αξία αλλά πώς να σας το πω, ε, η ποιότητα ας πούμε μπορεί να μην είναι ε, ο κεντρικός άξονας ε, της κατανομής τους. Εγώ νομίζω ότι εκεί θα υπάρξουν προβλήματα όπως και υπάρχουν, τα βλέπουμε. Άρα πρέπει να αλλάξει λίγο αυτή η τοποθέτηση. Ένα άλλο πρόβλημα είναι αυτό της συνοχής είσαστε εσείς, αλλά είναι και ο κύριος Κατάινεν για την μακροοικονομική υλοποίηση. Εγώ πολλές φορές ε, έχω κάνει ε, ε, έχω μιλήσει υπέρ κάποιων προγραμμάτων στην περιφέρειά μου και μάλιστα τα πένευα και τα ξαναπένευα και μετά μου είπανε όχι, όχι, όχι, μην λες τίποτα γιατί αυτά θεωρούνται δαπάνες και δεν είναι δυνατόν να τα εντάξουμε στα προγράμματα. Εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι στο νέο δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα αυτών των συνενώσεων. Ε, τα προγράμματα και οι συγχρηματοδοτήσεις από τη μία μεριά ε, να μην σημαίνουν από τη μεριά του κυρίου Κατάινεν ε, δαπάνη που δεν δικαιολογείται. Θα πρέπει να υπάρχει μια συνοχή και μια συνεκτικότητα και σε αυτή την ιδέα της συγχρηματοδότησης γιατί η ιδέα της συγχρηματοδότησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων είναι καλή και είναι και ελκυστική και βεβαίως μπορεί να υπάρχουν και σφάλματα, μπορεί να υπάρχουν και, και προβλήματα, αλλά τουλάχιστον να έχουμε κάποια στάση η οποία να είναι από την αρχή πιο συνεκτική και να υπάρχει δυνατότητα να ε, ε, προωθηθούν τα προγράμματα αυτά και να μην, να μην ε, υποχρεωνόμαστε μετά να κάνουμε επιστροφές και τα Θα πρέπει να βρούμε μία φόρμουλα, ένα τύπο, ώστε αυτή η συγχρηματοδότηση να μην, από τη δική σας την πλευρά, να μην υφίσταται μετά τις κυρώσεις της μακροοικονομικής αντιμετώπισης των δαπανών από τη μεριά του κυρίου Κατάινεν. Τέλος, όσον αφορά το ρόλο της ΕΤΕΠ. Έχετε δίκιο. Με κάποιο τρόπο θα πρέπει να βρούμε ε, ε, ε, ένα τρόπο να υπάρχει μεγαλύτερος έλεγχος από τη στιγμή που θα μπουν τα χρήματα στην ΕΤΕΠ. Θα πρέπει να βρεθεί λοιπόν ένας τύπος, ένας τρόπος όπου οι ευρωπαϊκοί κανόνες ε, είτε πρόκειται για την διευκόλυνση ε, για την Ευρώπη, είτε πρόκειται για οτιδήποτε άλλο. Ε, συγκεκριμένοι ευρωπαϊκοί κανόνες επί των οποίων έχουμε συμφωνήσει όλοι. Όταν τα χρήματα μπουν στην ΕΤΕΠ να μην εξαφανίζονται αυτοί οι κανόνες επειδή η ΕΤΕΠ δουλεύει με άλλη βάση ή με άλλους κανόνες και έχει εν πάση περιπτώσει μία αντιμετώπιση πολύ τραπεζική και πολύ συντηρητική γιατί ε, το πρόβλημα ε, είναι να μην μπορούν να ληφθούν υπόψη διάφοροι κανόνες από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έτσι ώστε να βοηθηθούν και προγράμματα τα οποία από καθαρά και αποκλειστικά τραπεζική σκοπιά μπορεί να είναι ε, άσχημα ή μπορεί να είναι επικίνδυνα, start-ups, νεοφυείς επιχειρήσεις. Αυτό που πρέπει να καταφέρουμε είναι η ΕΤΕΠ να έχει κανόνες τέτοιους και συνεργασίες με άλλες τράπεζες τέτοιες που ε, να ε, ε, δείξουν μια proactive στάση για το μέλλον. Και θα ήθελα και την άποψή σας για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαμε να επιτύχουμε αυτήν την διαφορετική αντιμετώπιση της ΕΤΕΠ. Ε, όχι μόνο τα καλά λόγια για την προπαγάνδα που κάναμε σε σχέση με το ΕΦΣΙ, αλλά ε, και ε, την αντιμετώπιση των νέων οικονομικών στοιχείων, της νέας οικονομίας, των νέων μορφών και, όχι μόνο, και που θα χρηματοδοτούνται και όχι μόνο να χρηματοδοτούνται οι πιο παραδοσιακές μορφές της πολιτικής. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω άλλο συνάδελφο να θέλει το λόγο. Ίσως θα πω κι εγώ κάτι λοιπόν. Και εγώ χαμογελώ όπως και εσείς. Ε, και συζητήθηκαν ε, πολλά θέματα σήμερα το πρωί. Uh, και νομίζω ότι και σε σχέση με τον Brexit είπατε ότι ε, ίσως προκύψει και μία τρύπα 15 δις λόγω του Brexit. Ακόμα βέβαια δεν ξέρουμε τι θέλει ακριβώς ε, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Ε, ε, ε, δεν ξέρουμε αν θα είναι ένα σκληρό Brexit και απλώς θα φύγουν ή αν θα είναι ένα υπιότερο και εν πάση περιπτώσει θα βρεθούν άλλοι τρόποι. Όμως χρειαζόμαστε και μια γρήγορη απόφαση από πλευρά της κυβερνήσεως του Ηνωμένου Βασιλείου. Οτιδήποτε και συμβεί βεβαίω, μέχρι να φύγει το Ηνωμένο Βασίλειο συνδέεται με επιδοτήσεις, κονδύλια, ευρωπαϊκά κτλ. Ερώτηση λοιπόν η Κομισιόν έχει ξεκινήσει κάποια εξειδικευμένη προσπάθεια έτσι ώστε να δει με ποιο τρόπο θα επιτηρούνται, ελέγχονται και ε, τα προγράμματα αυτά, ε, ε, τα επιδοτούμενα, πώς θα γίνεται ο οικονομικός έλεγχος, το auditing αυτών των κονδυλίων που έχουν δοθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και που θα δοθούν μέχρι τη στιγμή που θα φύγει. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, και Θέλω καταρχάς να επισημάνω ότι με τις επισκέψεις μου στα διάφορα κράτη-μέλη, με όλες τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια που συναντώ, προσπαθώ να ε, εξηγήσω στα κράτη, στα κοινοβούλια και τα 27 συνολικά. Την επόμενη εβδομάδα θα είμαι στην Ισπανία συγκεκριμένα για συναντηθώ με την ε, Ισπανική κυβέρνηση. Ποια είναι η κατάσταση τώρα, ποια είναι τα εργαλεία με τα οποία εργαζόμαστε. Είναι πολύ ενδιαφέρον και συναρπαστικό το θέμα αυτό και όντως κατά την προετοιμασία του προσεχούς δημοσιονομικού πλαισίου κάνουμε αυτή τη στιγμή εντατικέ συνομιλίε με του με τους επιτρόπου, του ε, επιτρόπου Γενικέ Διευθύνσει, στη δική μου Γενική Διεύθυνση. Εξετάζουμε δηλαδή ποια είναι τα καταλληλότερα δημοσιονομικά μέσα ή εργαλεία. Ξεκάθαρα δηλαδή, περισσότερα να καταφέρνουμε με λιγότερα μέσα. Αυτή είναι η... Αυτό λιγοτερα μεσα η αυτο ειναι το σύνθημα. Αλλά το perpetuum mobile δεν είναι εύκολο να βρεθεί το ακίνητο, όπως δεν μπορούμε και να τετραγωνίσουμε τον κύκλο. Πολλά είναι τα έργα, πολλά είναι, πολλές είναι οι περιφέρειες και τα κράτη που ζητούν, χρειάζονται χαμένες, ε, χαμένα κονδύλια, δηλαδή επιπλέον υποστήριξη και επιδοτήσεις. Ένας Γιώργος Φερρυπίν σε ένα ορεινό χωριό των Άλπαιων. Θέλει να αγοράσει ένα καινούριο γεωργικό μηχάνημα. Και πρέπει να δείξει την τράπεζα για να πάρει την επιδότηση του δανείου του ότι θα έχει την τόση επιδότηση από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό για την επόμενη επταετία με βάση την επιδότηση ανά εκτάριο. Ή έργα που η περιφέρεια θα μπορέσει να εκτελέσει επειδή έχει τη δυνατότητα να υποστηριχθεί, δεδομένου ότι ο προπολογισμό της περιφέρειας έχει ε, συμπιεστεί αρκετά, έχει υποστεί μεγάλε πιέσει, μόνο χάρη στην ευρωπαϊκή υποστήριξη. Επομένω, η Γεωργία, το Connecting Europe, ο, συνδέοντας την Ευρώπη, ορίζον 2020, η τα ποσά ή των, οι ενισχύσεις που θα χαθούν στο μέλλον, γενικά τα μετρητά το χρήμα, θα είναι το κύριο διακύβευμα. Και το ερώτημα βεβαίως, εάν έχει νόημα η συγχρηματοδότηση ή σε ποιο ύψος μπορεί αυτή να εξασφαλιστεί ή να είναι αποδεκτή. Στον πρώτο πυλώνα της γεωργικής πολιτικής, τις άμεσες ενισχύσεις. Είμαι πολύ επιφυλακτικός στην ιδέα των εθνικών χρηματοδοτήσεων. Έχει ανοίξει το θέμα μέσα από το έγγραφο αναλογισμού. Θα δοθούν οι απαντήσεις στις προτάσεις για το στο νομικό πλαίσιο το Μάιο. Ενώ στο δεύτερο πυλώνα υπάρχει περιθώριο σοβαρό για συγχρηματοδότηση σε μεγάλο βαθμό γιατί εκεί η περιφέρεια, ο εταίρος, επιδεικνύει και το δικό του το ενδιαφέρον, πόσο σοβαρά βλέπει, πόσο σημαντικό αξιολογεί, πόσο βιώσιμο κρίνει ένα ε, έργο. Δεν τραβάει δηλαδή απλώ χρήμα. Αναλαμβάνει και τη δική του την ευθύνη για την επιβεβαίωση, ε, για την επαλήθευση της ποιότητας. Το θέμα είναι αυτή η χρηματοδότηση θα είναι στο 20, στο 30, στο 40%. Θα πάει στην, ε, στο πρασίνισμα, θα μειωθεί στο 0. Θα ξανααυξηθεί σταδιακά μέσα από την ε, ποσόστοση την πολιετή της χρηματοδότησης. Το σχέδιο Juncker έχει τώρα μια ιστορια δυο δύο-τριών ετών και τη σχετική εμπειρία να μας προσφέρει. Θα συνεχίσει στις επόμενες την επόμενη δεκαετία. Και θα δούμε, και χρειάζεται εδώ πέρα μια ε, αξιολόγηση δαπανών, ένα spending review, γιατί δεν υπάρχει σχέδιο τόσο τέλειο που να μην χρειάζεται να αξιολογηθεί και να βελτιωθεί ύστερα από κάποια χρόνια υλοποίηση. Χαμένε ενισχύσει. Ή δάνεια από την άλλη. Grants ή loans. Και άλλη δυνατότητα διαχείριση. Τα grants ή ενισχύσεις είναι και μένα πάντα η ενισχυσει ειναι και μορφή χρηματοδότησης εγγυήσεις και δάνεια μπορούν να συμπληρώσουν σε, σε κάποιες περιπτώσεις να αντικαταστήσουν αλλά σε πολλές περιπτώσεις να συμπληρώσουν τις ενισχύσεις. Επίσης, ε, αναφερθήκατε στην ενίσχυση για startups, για νεοφυείς επιχειρήσεις. Για μένα, οι νεοφύση υπάρχονται στον ορίζοντα για την περίοδο μετά το 2020 πλέον. Στο κόσμο, επίσης, στην ε, στήριξη δηλαδή της θέσπισης, εγκαθίδρυσης και λειτουργίας στην αρχική φάση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και για μένα η νεοφύης επιχείρηση καθίσταται εταίρος στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και συμπληρωματικά μόνο εταίρος στο ΕΤΣΕ, στο νέο σχέδιο Juncker. Και βεβαίως οι νεοφύης θα πρέπει να είναι ικανές να ανταγωνιστούν τόσο τη Silicon Valley όσο και το Τελαβίβ ή το Σόρι. Και βεβαίως θα πρέπει οι νεοφύς επιχειρήσεις, startups να έχουν κάτι να προσφέρουν και για την ψηφιακή οικονομία. Γιατί έχουμε μετά τις startups, τις skylabs, τις unicorns, οι οποίες σε άλλες χώρες και περιοχές του κόσμου καθίστανται πιο ελκυστικές και άρα τραβούν περισσότερα κονδύλια και υποστήριξη. Η Βρετανία τέρη. είναι ακόμη μέλος το 2018 στον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, έχουν όλα τα καθήκοντα και τις ευθύνες που απορρέουν και τα δικαιώματα που απορρέουν από το γεγονός αυτό. Στην περίοδο μετά και μέχρι τα τέλη του 2020 συμμετέχουν πάλι με δικαιώματα και υποχρεώσει στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, παραμένουν δηλαδή εταίροι όσο είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα επόμενα χρόνια θα υπάρξουν έργα που θα υλοποιηθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επομένως, το 17, το 18 έχουμε αναλάβει ενδεχομένω κάποια υποχρέωση, έχουμε ε, προκηρύξει ένα έργο, έχουμε σχεδιάσει ένα έργο, έχει ξεκινήσει ένα έργο. Θα υλοποιηθεί αυτό, έχουμε δεσμευθεί. Και θα καταβάλουμε και τα σχετικά ποσά. Ακόμα και αν πρέπει η εκταμίευση να φτάσει μέχρι το 2023. Ο δε έλεγχος, η παρακολούθηση του έργου Τη εκτέλεσης του, της ανέγερσης κτλ. Ο έλεγχος ο δημοσιονομικός θα φτάσει και θα προχωρήσει και δικό σα καθήκον ω Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού, όπω και δικό μα ω Επιτροπή, όπω και του Ελεγκτικού Συνεδρίου αντίστοιχα ή του Συμβουλίου ΕΚΟΦΗΝ, θα είναι μια αρμοδιότητα και ένα καθήκον που ξεπερνά το έτος 2019. Έτσι αντιλαμβάνομαι εγώ το, δημοκρα... το παιχνίδι της δημοκρατίας, κανόνες δημοκρατικούς ελέγχω, τον, ε, την εκτέλεση των κονδυλίων που έχω πληρώσει. Είτε αυτά έχουν εκτελεστεί στο Λονδίνο, είτε στις Βρυξέλλες. Brexit. Ο πρόεδρος μου πριν από μερικές εβδομάδες είπε η πόρτα μένει ανοιχτή. Τα λάθη μπορούμε να τα διορθώσουμε. Αυτό ισχύει για μένα ως άνθρωπο, για μένα ως επίτροπο, ισχύει γενικότερα για την πολιτική και ένα δημοψήφισμα θα μπορούσε ακόμη να είναι ένα λάθος και μπορεί να διορθωθεί. Εάν τυχόν και γινόταν ένα δεύτερο δημοψήφισμα, αυτό είναι κάτι το οποίο αποφασίζει ο ευρωπαϊκός λαός, η Βουλή των Κοινοτήτων, η Πρωθυπουργό Τερέζα Μέη. Σας ευχαριστώ πολύ και βεβαίως είμαστε στη θέση σας για περαιτέρω επικοινωνία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ε, απαντήσεις σας. Θα δώσω ξανά το λόγο στον εισηγητή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ντέρεκ. Ευχαριστώ και τον Επίτροπο για τις ε, παρατηρήσεις του και για τις ε, θέσεις του. Δυστυχώς, ε, εκεί που κάθεται να του γυρίζω την πλάτη, δεν είναι θέμα ευγένειας. Πολλά από αυτά τα οποία είπατε Νομίζω ότι βρίσκουν σύμφωνο εμένα και αρκετούς συναδέλφους και νομίζω η Επιτροπή μας και το Κοινοβούλιο συνολικά θέλει να ακολουθήσει αυτά τα οποία είπατε. Ξανά τώρα για την πολιτική συνοχή. Μιλήσατε για το νησιν 2, νησιν 3. Υπήρχαν νομίζω διαφορετικά προβλήματα στην διαδικασία κατάρτισης των νέων περίοδων και βεβαίως ε, αν είχαν συμφωνήσει η Κομισιόν και η Κοινοβούλιο το 2012 πριν την αρχή της νέας προγραμματικής περίοδου για την ε, νομική βάση της ε, πολιτικής συνοχής, τότε οι διαπραγματεύσεις του τριμερούς διαλόγου που κράτησαν τρεις προεδρίες για την οριστική απόφαση θα είχαν ολοκληρωθεί πολύ πιο γρήγορα γιατί ολοκληρώθηκαν τελικά άνοιξη του 2014 και είχαμε κάποιες ε, μεθόδους που υποτίθεται ότι θα ήταν καινοτόμες, κάτι το οποίο ακούγονταν καλό, αλλά τελικά είχαμε ακόμη μεγαλύτερες ε, καθυστερήσεις και οι εταιρικέ συμφωνίες μεταξύ Κομισιών και κρατών μελών, ε, άλλο ένα νέο στοιχείο οδήγησε σε άλλη μια καθυστέρηση 1,5 έτους και σήμερα βλέπουμε ότι δεν αξίζουν ούτε το χαρτί στο οποίο γράφτηκαν. Και μετά από αυτές τις ε, συμφωνίες ε, μπόρεσαν να ξεκινήσουν τα επιχειρησιακά προγράμματα. Άλλος ένας χρόνος χάθηκε. Ο συνάλφος και επίσης έθεσε το ζήτημα της εξάντερεσιμότητας ε, που θα πρέπει να εξεταστεί. Βεβαίω αυτό ήταν μια καλή πρόθεση, αλλά τελικά στην εφαρμογή οδήγησε σε αυξημένη γραφειοκρατία και θα πρέπει νομίζω να ξανασκεφτούμε σε ποιο βαθμό ήταν αποτελεσματικές οι διαδικασίες μας, δηλαδή αν επιτευχθεί ο σκοπός για τον οποίο ε, τις υιοθετήσαμε. Βεβαίω ναι, επιχορήγηση, δάνεια, εγγυήσει ε, είναι ένα θέμα νομίζω ότι στην ε, πολιτική έρευνας ε, μόνο με επιδοτήσεις μπορούν να εργαστούν και πρέπει να γνωρίσουμε ότι έχουν δικαίωμα και στο σφάλμα βέβαια και σε πολλά ζητήματα πολιτικής συνοχής έχουν έτσι τα πράγματα και βέβαιω ισχύει και το ότι αυτό το οποίο δεν κοστίζει τίποτα δεν αξίζει και τίποτα και επίσης συχνά διαπιστώνουμε πως τα κριτήρια μας όταν πάμε στην ε, εφαρμογή ε, συγκρούονται με τα κριτήρια επιδοτήσεων και Έχουμε δηλαδή πολύ διαφορετικές ε, διατάξεις, οι οποίες μάλιστα είναι αλληλοαποκλειόμενες. Έχουμε και μια άλλη έκθεση την οποία θα ήθελα να αναφέρω. Είναι οι ειδικέ εκθέσεις του ελεγκτικού συνεδρίου που έχουν γίνει μία έκθεση. Οι έκθεση ε, αυτές για εμένα και για πολλούς ε, συναδέλφους είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για να δούμε τις λεπτομέρειες ε, της ευρωπαϊκής ε, πολιτικής και μας ε, δίνουν χρήσιμες πληροφορίες που βεβαίως αφορούν και τις εκθέσεις απαλλαγής. Αλλά αυτό θα το δούμε σε εκείνη την έκθεση. Για μένα ιδιαίτερη σημασία είχε η έκθεση για την βοήθεια στην Ουκρανία όπου υπάρχουν διάφορες ελλείψεις, ότι θα πρέπει να φανούν περισσότερο οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να συνδεθούν περισσότερο με την Ουκρανική κυβέρνηση, ότι η Ουκρανία θα πρέπει να προχωρήσει σε ένα σύστημα αποτελεσματικής φορολογίας ε, για να μην μένουν εκτός οι ολιγάρχες ε, και βεβαίως και ο ε, οργανισμός αυτός ο οποίος ιδρύθηκε και με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της ε, διαφθοράς ε, αντιμετωπίζει δυσκολίες στην Ουκρανία και πρέπει να στηριχθεί και πρέπει να ελεγχθεί επίσης περισσότερο ο τραπεζικός τομέας στην Ουκρανία για να εμποδιστούν αυτές οι μεγάλες εκροές κεφαλαίων που έχουν ε, διαπιστωθεί γιατί τα χρειάζεται αυτά τα χρήματα η χώρα. Για τον έλεγχο της αλληλείας βλέπουμε πως πολλά θέματα ε, δεν πολλές διατάξεις δεν εφαρμόζονται στα κράτη-μέλη, στα θέματα αλληλείας και συχνά έχουμε είτε ωρεοποιημένα είτε λανθασμένα δεδομένα με τα οποία εργαζόμαστε και λείπουν επίσης αρκετά δεδομένα και η βοήθεια επίσης ε, για τα Δυτικά Βαλκάνια η εκεί και αυτή έχει αρκετές ελλείψεις ε, και βεβαίως και το καταπίστευμα αυτό για την ε, Αφρική ξεκίνησε οπωσδήποτε ως κάτι το οποίο είχε καλές προθέσεις και τα κράτη-μέλη τα οποία θα ήθελαν να εμπλακούν όμως ε, περισσότερο δεν είχαν αυτή την ευκαιρία. Οι δε πληρωμές που ελπίζαμε ότι θα έρθουν από τρίτα μέρη δεν ήρθαν και το διοικητικό κόστος επίσης ε, ε, δεν είναι τόσο λογικό σε σχέση με, την, με το συνολικό ύψος της χρηματοδότησης. Και πρέπει βεβαίω να έχουμε και έναν προσανατολισμό με τους γενικότερους στόχους της αναπτυξιακής πολιτικής. Αυτά τα ολίγα για τις ειδικέ εκθέσεις του ελεγκτικού συνεδρίου. Σας ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση και αναμένω βεβαίως τις ε, τροπολογίες των ε, συναδέλφων για να καταλήξουμε στην τελική μορφή της έκθεσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, κύριε Σιγητά και βεβαίως να ευχαριστήσω και τον κύριο Επίτροπο που ήρθε ξανά μαζί μας και θα σας διασφαλίσουμε ένα μπάτζ για να μπαίνετε όποτε θέλετε και όπως θέλετε στο Κοινοβούλιο. Επόμενο θέμα αφορά την ανανέωση του ελεγκτικού συνεδρίου. Δύο λεπτάκια διακόπτουμε έτσι ώστε να εγκαταλείψουν την αίθουσα όσοι πρέπει να φύγουν. Okay, colleagues, we can... Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορούμε να ξαναρχίσουμε στο 48 τώρα τη ημερήσια διάταξη. Μερική ανανέωση των μελών του ελεγκτικού συνεδρίου. Υποψήφια από το Βέλγιο. Κυρία Τόρτλμπουμ είναι εδώ παρούσα. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Θα σας καλέσουμε να κάνετε την πεντάλεπτη σα παρουσίαση και μετά ο εισηγητής θα λάβει το λόγο. Παρακαλώ κύριε Τέρτελμπλουμ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε εισηγητά, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι. Μεγάλη χαρά και τιμή ε, ε, αισθάνομαι που βρίσκομαι ενώπιόν σας σήμερα ως υποψήφιο μέλος ε, του Ελεκτικού Συνεδρίου ε, ε, προτινόμενη από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση του Βελγίου. Έχω σπουδάσει οικονομικά και διοίκηση επιχειρήσεων και πρόκειται για ενασχόληση την οποία στην Λουβέν ως καθηγήτρια πανεπιστημίου έχω ε, βελτιώσει. Έχω υπάρξει πολλές φορές αναπληρώτρια υπουργό, καθώς επίσης ε, και υπουργό στην Φλάνδρα. Επίσης ε, έχω υπάρξει επι, υπεύθυνη για, την, ε, για τους δημόσιους λογαριασμούς και επίσης Ήλεξα τους προϋπολογισμούς του 2014 και του 2015, καθώς επίσης ε, και την υλοποίηση του συστήματος ελέγχου των λογαριασμών ε, του Ευρωπαϊκού Προτύπου από την ε, κυβέρνηση της Φλάνδρας. Επίσης, έχω περάσει από τρία υπουργεία που αφορούν το άσυλο και την μετανάστευση, καθώς επίσης και το Υπουργείο των Εσωτερικών. Κάθε φορά, σε οποιαδήποτε θέση, έχω προσπαθήσει ε, να συνεργαστώ στενά ε, με ελεγκτικούς οργανισμούς Έχω ζητήσει ελέγχους από το ε, Συμβούλιο ε, του Βελγίου που είναι παρόμοιο με το ελεγκτικό συνέδριο ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω συνεργαστεί ε, επίσης με την Standing Police Monitoring Committee, επίσης με την Επιτροπή Αναθεώρησης του Βελγίου, καθώς επίσης και με την ε, ανεξάρτητη αρχή ελέγχου εσωτερικών πληροφοριών και δικαιοσύνης. Έχω δουλέψει ε, και σε αυτή την περίπτωση με ε, Ευρωπαίους αξιωματούχους. Επίσης, για έξι χρόνια από την θέση μου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης έχω εργαστεί με Ευρωπαίους συναδέλφους στα πλαίσια του Συμβουλίου Δικαιοσύνης. Αυτά τα έξι χρόνια η ε, αποτέλεσαν μεγάλη πρόκληση αλλά ε, μου έδωσαν και μεγάλη συνάφεια όσον αφορά ε, τα ευρωπαϊκά θέματα. Επίσης ε, ε, είχα την δυνατότητα να συνεχίσω την ακαδημαϊκή μου καριέρα, ε, να αναφερθώ σε θέματα που αφορούν το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να έρθω σε επαφή με ανθρώπους προερχόμενους από όλο τον κόσμο και επομένως να συμβάλλω θετικά την εξέλιξη, με συγγνώμη και αυτή η διαδικασία θετικά στην εξέλιξη της καριέρας μου. Η συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κυρίως δε με την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, θεωρώ ότι το ελεγκτικό συνέδριο προσυπογράφει την, στην ανάγκη δημοκρατικής ε, λογοδοσίας. Ε, ε, εάν οριστώ στη θέση αυτή, θα συμμορφωθώ πλήρως στις απαιτήσει της θέσης. Θα, θα δείξω ακαιρεότητα και αμεροληκτικότητα ψία. Ε, ε, δεν πρόκειται να, να, να ε, πάρω οδηγίε από οποιονδήποτε, οποιαδήποτε κυβέρνηση ή θεσμό. Είμαι πεπισμένη ε, ότι ε, οι διαφορετικές προσεγγίσεις, ε, τα διαφορετικά βιογραφικά και η πολυμορφία, καθώς επίσης και η ισορροπία των φύλων είναι θέματα πολύ θετικά. Θεωρώ ότι η επερχόμενη περίοδος είναι σημαντική και για το Ελεκτικό Συνέδριο και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μπροστά μας μας περιμένουν πολύ σημαντικές αποφάσεις, σημαντικές πολιτικές για την Ευρωπαϊκή Ένωση, εργαλεία χρηματοδότηση, και επομένω και εξέλιξη του ελεγκτικού συνεδρίου. Ωστόσο αυτές τι διαδικασίε θα μπορούσαμε να τι δούμε σαν πρόκληση για το ελεγκτικό συνέδριο εάν ε, ε, έχω θετική γνωμοδότηση από τη δικιά σας ε, πλευρά θα προσπαθήσω να αντιμετωπίσω αυτές τις προκλήσεις έτσι ώστε να τις μετατρέψω σε ευκαιρίες. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και αναμένω τα σχόλιά σας. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Οι Βέλγοι εξοφίσιο θεωρούνται Ευρωπαίοι. Παρακαλώ, εισηγητής, κύριε Τάραντ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι και θεωρώ ότι είναι τιμή μου που είμαι εισηγητής για τον ορισμό ενός νέου μέλου στο ελεγκτικό συνέδριο προερχόμενου από το Βέλγιο μετά από, μετά από πρόταση της ε, κυβέρνησης του Βελγίου γιατί βελτιώνει την ισορροπία των φίλων στο ελεγκτικό συνέδριο ε, και μπορεί να αποτελέσει και ε, καλή απάντηση του βελγικού, της βελγικής κυβέρνησης με τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίσαμε με το προηγούμενο υποψήφιο. Έχω μία ερώτηση μονάχα προς την υποψηφία. Εάν ε, κάποιος έχει μελετήσει οικονομικά και μετά από αυτό ε, ε, τα δίδαξε τα οικονομικά σε άλλους, θεωρώ τεκμέρο ότι αυτό αποτελεί θετικό στοιχείο γιατί ε, τα οικονομικά είναι μεγάλο κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οπωσδήποτε ε, ε, πρέπει να υπάρχει αμεροληψία και χωρίς προκατάληψη οικονομικός έλεγχος σε όλες τις χώρες. Η ερώτησή μου λοιπόν προέρχεται από την γραπτή σας απάντηση στην ερώτηση 13. εκεί όπου προσπαθούμε να μάθουμε την στάση που έχετε στη δική σας χώρα. Αλλά ακόμα πιο σημαντική είναι η στάση σας προς άλλες μικρές χώρες, όπως η Εστονία ας πούμε. Και σας ρωτώ, εάν πληροφορηθείτε ότι η ε, ε, ε, η υπηρεσία πρόθεσης των επιχειρήσεων στην ε, Εστονία έχει εγκρίνει ας πούμε να ανοίξει στη Μαλαισία ε, γραφείο από επιχείρηση που δεν υπάρχει. Θα δώσετε απαλλαγή ή όχι. Κύριε όπως ε, είπα και προηγουμένως, η ανεξαρτησία και η αμεροληψία ε, θα πρέπει να είναι αδιαμφισβήτητες και αδιαπραγμάτευτες ε, για οποιονδήποτε θέλει ε, να ενταχθεί στο ελεκτικό συνέδριο. Θα πρέπει να γίνει οπωσδήποτε οικονομικός έλεγχος. Βεβαίως εγώ δεν θα κάνω καμία διαφοροποίηση μεταξύ χωρών. Δεν πρόκειται να λάβω οδηγίες για οποιαδήποτε χώρα ή από οποιαδήποτε χώρα. Εάν και εφόσον υπάρχει κάποια ατασταλία, εάν και εφόσον προκύψει απάτη θα, θα αναλάβει το θέμα η Όλαφ. Η Όλαφ λοιπόν εάν παραστεί ανάγκη θα ξεκινήσει, ε, ε, θα αρχίσει να διαρευνά την ε, υπόθεση Νομίζω ότι οποιαδήποτε χώρα, μικρή, μεσαία, μεγάλη, ε, χώρα που βρίσκεται στο κέντρο της Ευρώπης ή στην περιφέρεια της Ευρώπης θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο γιατί αν ε, ε, κάποιος πραγματικά θέλει να γίνει μέλος και μέρος του ελεγκτικού συνεδρίου αυτή είναι μία εκ των ουκάνευ αρχή. Ευχαριστώ ο κύριος Στοιχόφσκι. Πρόεδρε, ευχαριστώ με διπλή ιδιότητα είμαι εδώ. Θα ήθελα λοιπόν να σας δώσω καταρχάς ε, τις ερωτήσεις του κυρίου Σάουαρμα, ο οποίος ε, είναι συντονιστής εκ μέρους του ΕΛΚ, δεν μπόρεσε όμως λόγω πολύ σοβαρών υποχρεώσεων στην πατρίδα του να έρθει εδώ σήμερα και μετά θα ακολουθήσουν δικές μου ερωτήσεις εκ μέρους του κυρίου Σαρβάμα λοιπόν. πώς θα, συνεχί... πώς θα βελτιώσετε, πώς θα συμβάλλετε στην περαιτέρω βελτίωση του έργου του Ελεκτικού Συνεδρίου και δική σας δουλειά ως μέλος του Ελεκτικού Συνεδρίου ε, στη μελλοντική σας εντολή, πώς θεωρείτε ότι πρέπει να αναπτυχθεί και αν ήταν να, να κάνετε μια επιλογή μεταξύ τομέων στους οποίους θα έπρεπε να επικεντρώσει το ενδιαφέρον του το Ελεκτικό Συνέδριο, ποιοι θα ήταν αυτοί. Επίσης από τη δική μου την ερώτηση, στην τσεχική γλώσσα αυτή τη φορά. Και χωρίς μικρόφωνο. Εδώ χαιρόμαστε που σας βλέπουμε ως υποψήφια. γιατί χαιρόμαστε να έχουμε υποψηφίους για τους οποίους δεν υπάρχουν υπενιγμοί ή κατηγορίες που διερευνά ή όλαφ. Καλό λοιπόν αυτό. Πρώτον και δεύτερον, χαίρομαι γιατί βλέπω ότι είστε και ενθουσιώδης τύπος. Βλέπω από βίντεο που έχω βρει στο ίντερνετ ε, για εσάς ότι είστε πολύ ενθουσιώδης τύπος και ε, ενδιαφέρομαι, ε, με, χαροποιεί αυτό. Ωστόσο το ελεκτικό συνέδριο είναι ένα βαρετό όργανο, μια βαρετή ζωή. Όλο αυτό τον ενθουσιασμό, την ενέργειά σας, πώς θα την συγκεράσετε με τις δραστηριότητες, τις βαρετές αυτές δραστηριότητες ενός δημοσιονομικού ελεγκτή. Και θα είσαστε τελικά μαύρο πρόβατο ή άσπρο πρόβατο. Η απάντηση, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Αν κοιτάξουμε στο μέλλον του συνεδρίου, και στα σημεία που θα πρέπει να δώσουμε περισσότερη έμφαση. Αυτή τη στιγμή η Επιτροπή εξετάζει τον προπολογισμό περισσότερο στοχευόντας σε αποτελέσματα. Νομίζω ότι εκεί έχει τοποθετηθεί το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αντίστοιχα και του ελεγκτικού συνεδρίου πρέπει να αλλάξει ο τρόπος εργασίας. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ των ελέγχων που έχουν να κάνουν με τη συμμόρφωση αφενός και τα αποτελέσματα αφετέρου, αλλά πιστεύω ότι και ο Πρόεδρος και τα λοιπά μέλη τίνουν περισσότερο προς τον έλεγχο με βάση την αποδοτικότητα, γιατί μπορεί κανείς να βρει ε, στοιχεία, ε, έργα τα οποία είναι επωφελή για τον πολίτη. Ταυτόχρονα τρία τα τρία ε, efficiency, effectiveness και economy, πρέπει να συνδυάζονται, δηλαδή αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και οικονομία για να κερδίσουμε και την ε, εμπιστοσύνη του Ευρωπαίου πολίτη στα ευρωπαϊκά όργανα, στο ευρωπαϊκό όραμα. Ιδιαίτερος λοιπόν καλωσορίζω την ε, διάθεση για περισσότερη ε, αξιολόγηση των δημοσιονομικών με βάση την αποδοτικότητα των έργων, γιατί εκεί ε, αποδεικνύεται και η ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία. Ταυτόχρονα θα ήθελε και περισσότερη επικοινωνιακή, πιο αποτελεσματική, επικοδο... Ε, ε, αποτελεσματική πολιτική. Χαίρομαι που το ελεκτικό συνέδριο και η έκθεσή του για το 2016 δημοσιοποιήθηκε στα κράτη-μέλη και έτσι έγινε η συζήτηση και όχι μόνο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και με άλλους εμπλεκόμενους φορείς. Χαίρομαι λοιπόν και πιστεύω ότι θα πρέπει να συζητούμε τα θέματα που έχουν μεγαλύτερη απήχηση και ε, κερδίσουν το ενδιαφέρον του πολίτη. Ταυτόχρονα και στην επόμενη έκθεση βλέπετε ότι υπάρχει μεγαλύτερη έμφαση στα θέματα της μετανάστευσης, ε, της ασφάλειας, θέματα που διατηρούν τη σημασία τους όπως και τη προσθέμενη αξία τη Ευρώπη. Επίση, η προσθέμενη αξία ε, πρέπει να αποδεικνύεται, πρέπει να αποδεικνύεται ότι τα λεφτά του Ευρωπαίου φορολογούμενου δαπανώνται σωστά. Για την ενεργειά μου και την ενεργητικότητα μπορώ να επιδείξω. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να προσφέρω με αυτήν, να συμβάλλω στη δουλειά του ελεγκτικού συνεδρίου. Ξεκίνησα λέγοντα ότι ήμουνα για δύο χρόνια υπουργό ε, ε, Εθνικής Οικονομίας και Δημοσιονομικών και ω εκ τούτου είχα να κάνω με το ελεγκτικό συνεδρίο το βελγικό. Ταυτόχρονα ήμουν και υπουργό εταιρικών με θέματα μετανάστευση και προσφυγικά και με θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχω συνεργαστεί. Ε, μπορώ να σα δώσω παράδειγμα σε σχέση με το τι μπορεί να προσφέρει ένα ελεκτικό συνέδριο. Είχαμε μια έκθεση ειδική από το Ευρωελγικό Ελεκτικό Συνέδριο όταν ήμουν στην κυβέρνηση για τον υπερπληθυσμό στι φυλακέ. Ε, έγινε ένα master plan, αλλά περάσανε πέντε χρόνια και ακόμα συζητούσαμε το σχετικό αυτό, τη σχετική έκθεση δηλαδή, στο, ε, η βελγική κυβέρνηση. Επίσης έχω εμπειρία από το Συμβούλιο. Έξι χρόνια ήμουνα μέλος του Συμβουλίου ε, των Ιστορικών και της Δικαιοσύνης. Πιστεύω ότι με αυτά μπορώ να προσφέρω. Κυρία Γελασέντερ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε κυρία Τουρτολμπούμ στην Επιτροπή μας. Πρώτα απ' όλα. Και εγώ θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου γιατί ε, κερδίσαμε ε, όσον αφορά ε, την ισορροπία των φίλων με τη δική σας υποψηφιότητα. Αυτό είναι θετικό. Επίσης βλέπουμε ότι είχατε και θέσεις οι οποίες ε, δεν είχαν καλυφθεί μέχρι τότε από γυναίκες όπως ας πούμε Υπουργείο Εσωτερικών Δικαιοσύνης και λοιπά στη χώρα σας στο Βέλγιο. Και αυτό είναι πολύ καλό. Χαίρομαι λοιπόν γι' αυτό. Βλέπω το βιογραφικό σας, είναι πολιτική η διαδρομή σας και είναι γεγονός ότι και εμείς ε, Γνωρίζουμε πολύ καλά ε, την ε, πολιτική και στο Βέλγιο έχει ιδιαίτερη σημασία. Επίσης, ε, σημαντική η σχέση σας με τον κύριο Πίνστεν. Και ίσως θα μπορούσατε να μας πείτε πότε προτίθεστε να εγκαταλείψετε όλες τις ε, πολιτικές θέσεις οι οποίες κατέχετε σε περίπτωση που προχωρήσει θετικά ε, η υποψηφιότητά σας, ε, έτσι ώστε να ασχοληθείτε με το ελεγκτικό συνέδριο. Δεύτερον, στο βιογραφικό σας βλέπουμε ότι είσαστε γυναίκα με πολύ συγκεκριμένες και ισχυρές ε, πεπιθήσεις, τις οποίες ε, ε, υλοποιείτε έτσι με πολύ μπρίο, αλλά είναι γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν εκφραστεί επικρίσεις όσον αφορά μελλοντικές πολιτικές της Ευρώπης, όπως ας πούμε για την μετανάστευση. Εγώ μίλησα βέβαια ε, και με την ε, κυρία ε, Αρενά για τα θέματα αυτά και έχω διαβάσει και τον τύπο αυτό που χρειαζόμαστε στο ελεγκτικό συνέδριο είναι μία ε, ομάδα, ε, δηλαδή να μπορέσουν τα μέλη του ελεγκτικού συνεδρίου να λειτουργήσουν σαν ομάδα, γιατί μπαίνουμε σε μία νέα εποχή, μπαίνουμε σε ύδατα, ε, αν όχι αχαρτογράφητα, αλλά εν πάση περιπτώσει περίπλοκα και επομένως χρειαζόμαστε ένα ελεγκτικό συνέδριο που να μπορεί να συνδιαλέγεται, που να μπορεί να συζητά και να λειτουργεί σαν ομάδα. Τέλος, βλέπω ότι το 2016 ασχοληθήκατε και με την ενεργειακή μετάβαση, όμως θα μπορούσατε να μας πείτε δύο, δύο λόγια γι' αυτό. Και βέβαια, διαβάζοντα και ακριβώ πώ αντιμετωπίσατε τα θέματα αυτά και σε σχέση με τι ΗΠΑ, βλέπω ότι είσαστε ε, γυναίκα με έντονε πεπιθήσει. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτησή σας. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω με το εξισή πολιτική μου εντολή, να μου την δώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την στήριξή του, προφανώς θα παρετηθώ από όλες μου τις ε, θέσεις. Αυτή τη στιγμή είμαι μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου της Αμβέρσας, είμαι βουλευτής στο Βελγικό Κοινοβούλιο και μέλος ε, των φίλων του Μουσείου Μόδας και από εκεί θα παρετηθώ γιατί υπάρχει βεβαίως και η Επιτροπή Ιδεοντολογίας και αν κάποια στιγμή μπορούμε να το συνδυάσουμε με κάτι, κάποια φιλανθρωπική δραστηριότητα θα μπορούσα να ρωτήσω την Επιτροπή Ιδεοντολογίας εάν επιτρέπεται ή όχι αλλά για να ξεκινήσω να κάνω μια νέα αρχή θα παρετηθώ από τα πάντα. Ό, δεν είναι δύσκολο, θα γράψω μια επιστολή και θα πω από αύριο παρετούμε και θα βρουν κάποιον άλλον. Νομίζω να είναι κάποιο πρόβλημα και νομίζω ότι στο κοινοβούλιο έχουμε τη σχετική εμπειρία και είναι κάτι το φυσιολογικό. Και είναι φυσιολογικό γιατί η ανεξαρτησία πρέπει να μην αμφισβητείται. Αν κάποιος είναι ανεξάρτητος δεν μπορεί να έχει και άλλες ε, δραστηριότητες που δεν είναι σαφές ε, εάν είναι ανεξάρτητος κατόπιν για την παρέτησή μου. Κάποια στιγμή στο Βέλγιο δίναμε επιδοτήσεις για ηλιακά πάνελ και ανεμογεννήτριες ε, σε σπίτια, σε ιδιωτικές εταιρείες. Είχε ξεκινήσει αυτό το πρόγραμμα το 2001, αλλά χρειάστηκε να φτάσουμε μέχρι το 2014 για να γίνει μία ανάλυση σε βάθος για το τι σημαίνει αυτό σε βάθος χρόνου και για τους λογαριασμούς σπιτιών και εταιριών. Έπρεπε λοιπόν να βρεθεί μια λύση, το αποφάσισε και η πλειοψηφία. βρήκα μια λύση, αλλά μετά το ζήτημα προσωποποιήθηκε και ήμουν υπουργό ε, για 8 χρόνια και όλοι ξέρουμε βεβαίως πόσο παρεμβαίνει η πολιτική ζωή στα προσωπικά μας και αν γίνουν τα πράγματα τόσο προσωπικά ώστε δεν μπορούμε πλέον να σκεφτούμε αντικειμενικά ε, και όπως είχαν γίνει αποφάσισα τότε να παρετηθώ και ανέκτησα την ελευθερία λόγου μου και είχα και την ευκαιρία να σπουδάσω και ένα εξάμεινο στο Γέιλ. Όσον αφορά την ισορροπία των φίλων, γιατί και αυτό αναφέρθηκε, ε, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ θετικό το ότι το ελεγκτικό συνέδριο ξεκαθαρίζει το θέμα αυτό γιατί εγώ ε, αν στηρίξετε θα έχουμε μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ των μελών του ελεγκτικού συνεδρίου αλλά υπάρχει ένας ολόκληρος οργανισμός και πρέπει να γνωρίζουμε ακριβώς την ισορροπία των φίλων στο σύνολο του οργανισμού. Εγώ πάντα απέδιδα μεγάλη σημασία σε αυτό, γιατί όταν ήμουν υπουργό Εσωτερικών ε, ζήτησα να γίνει έλεγχος ε, στην Ομοσπονδιακή Αστυνομία του Βελγίου, γιατί ήταν ένα ανδροκρατούμενο περιβάλλον και οι γυναίκες ήταν πιο χαμηλόβαθμες, οπότε ε, θα το δω αυτό το ζήτημα και θα στηρίξω οποιονδήποτε άνδρα ή γυναίκα στις φιλοδοξίες του Βεβαίω, όταν μιλάμε για αξιολόγηση, η σημασία έχει να είναι ο καλύτερο ή η καλύτερη. Οπότε θα παρακολουθήσουμε αυτό το σύστημα. Υπάρχει και μια ετήσια έκθεση, αλλά θα το δούμε στο σύνολο του οργανισμού του ελεγκτικού συνεδρίου. Σας ευχαριστώ κυρία Λαμπάγεβα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε ανεμή στην Επιτροπή μα. Νομίζω πω η εμπειρία σα. Ε, και η ενέργειά σας ε, θα φέρει μια νέα προοπτική στο ελεγκτικό συνεδρίο και στην Επιτροπή μας ε, και προσωπικά το αναμένω αυτό με ανυπομονησία. Εργαστήκατε σε δύσκολα ζητήματα στο Βέλγιο. Το Βέλγιο είναι και αυτό μια δύσκολη χώρα και νομίζω ότι θα είστε πάρα πολύ καλοί στα περίπλοκα θέματα. Θα σας εξηγήσω τη διαφορά ανάμεσα στα περίπλοκα και τα πολύπλοκα. Ε, λοιπόν, υπάρχει, όπως είπαμε, ένας περίπλοκος ε, προϋπολογισμός ε, και χαίρομαι που αναφέρατε ακριβώς τον έλεγχο με βάση την απόδοση, την προστιθέμενη αξία και χαίρομαι γιατί έχετε την εμπειρία και από την εθνική σκοπιά και από την ευρωπαϊκή πτυχή. Αναφέρατε επίσης τη μεγάλη σημασία του να δίνουν τα κράτη-μέλη ακριβή πληροφορίε στην Κομισιόν γιατί δεν μπορεί το ελεγκτικό συνέδριο να ζητήσει απευθεία στοιχεία. Θα ήθελα λοιπόν να σα ρωτήσω. Ε, θα έπρεπε το ελεγκτικό συνέδριο να έχει την δυνατότητα να ζητάει απευθεία από τα κράτη-μέλη πληροφορίε. ή θα θέλετε να διατηρηθεί το status quo και να υπάρχει δυνατότητα να ζητήσουν πληροφορίε μόνο μέσω της ε, Κομισιόν και εφόσον έχετε δει και τις δύο πτυχές, ποια είναι η άποψή σας. Σας ευχαριστώ. Σωστές ε, πληροφορίες ε, είναι, αποτελούν τη βάση την, του σωστού οικονομικού ελέγχου. Auditing σημαίνει έλεγχους της ε, σωστής δαπάνης ε, των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Επομένως, νομίζω ότι πρώτα πρέπει να έχει κανείς πληροφόρηση από την Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή. Βεβαίως και με εθνικές τοπικές αρχές, δήμους, κοινότητες κλπ. Πάντως πιστεύω ότι πρώτα πρέπει να στρέφεται κανείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να έχει αξιόπιστες πληροφορίες. Εάν πάει κανείς απευθείας ε, στο ε, κράτος μέλος ε, θα πρέπει να είναι κανείς βέβαιος απόλυτα για την νομική διαδικασία γιατί ούτως ή άλλως πρέπει να ε, ετοιμάζεται η έκθεση και να δίνεται και η δυνατότητα ε, σχολείων. Ε, γι' αυτό με βλέπετε επιφυλακτική στο να πηγαίνει κανείς απευθείας να στρέφεται προς τις χώρες μέλη. Πιστεύω ότι πρώτα στρέφεται κανείς στην Κομισιόν. Ναι, είναι γεγονός ότι μπορεί να παραμείνουν κάποιες γκρίζες ζώνες και επομένως να χρειάζεται κανείς επιπλέον πληροφορίες από την χώρα μέλος. Το πρώτο πιστεύω είναι συνεργασία ε, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά βεβαίως δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει σε κάποια περίπτωση να πάει απευθεία στο κράτος μέλος. Ο κύριος Φλάναγκαν. Ευχαριστώ πολύ. Ένα θετικό σκέλος της, ε, του, της υποψηφιότητάς σας ε, ε, είναι ότι πραγματικά βοηθά την ισορροπία των ε, φύλων. Αλλά για να επιστρέψουμε στο θέμα της παρέτησής σας ε, σε σχέση με το θέμα που είπατε. Είναι γιατί από ό,τι έμαθα, μάθατε ότι ο φόρος ήταν αντισυνταγματικός, γιατί ο φόρος υπήρχε ήδη και Κοιτάξτε, ε, εσείς στη νέα σας θέση θα κληθείτε να ελέγχετε την νομιμότητα ε, της ε, χρήσης των πόρων. Δεύτερον, ποια είναι η άποψή σας όσον αφορά την παρανόηση Ε, ε, ανάμεσα από τον διπλό ε, έλεγχο ενώ μπορεί να γίνει ένας ενιαίος έλεγχος εάν τα πράγματα είναι καλά γίνεται ο έλεγχος και βγαίνει το αποτέλεσμα τρίτον όσον αφορά τους λογαριασμούς ή ε, ε, διορθώσεις ε, μπορεί να γίνουν μονάχα σε την εκδοχή του ελεγκτικού συνεδρίου και όχι στους αρχικούς λογαριασμούς. Ευχαριστώ πολύ, λέει η κυρία Μπλουμ. κοιτάξτε, όταν μια κυβέρνηση πάρει μια απόφαση, το δικαστήριο μπορεί να ανακαλέσει κάποιες διαδικασίες. Έτσι είναι οι διαδικασίες, έχουμε ανεξάρτητη δικαιοσύνη συνέβη και στη δικιά μου περίπτωση αλλά και σε άλλες περιπτώσεις και μετά η κυβέρνηση καλείται να πάρει μια άλλη απόφαση. Είναι post factum ανάλυσης. Την κάνουν αυτήν την ανάλυση λοιπόν, ε, όχι μόνο στη δικιά μας περίπτωση αλλά και σε άλλες. Δεύτερον, ναι βεβαίως είμαι πολιτικός ε, αλλά είμαι πεπισμένη ότι ε, διαφορετικά προφίλ και επαγγελματικέ εμπειρίες μπορούν να εμπλουτίσουν το ελεκτικό συνέδριο. Βλέπω ότι τα μέλη του ελεκτικού συνεδρίου προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από Εθνική Διακυβέρνηση, ε, Συμβούλιο Υπουργών, αλλά υπάρχουν και τεχνοκράτες, υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν ακαδημαϊκό ε, υπόβαθρο. Ε, το Ελληνικό Συνέδριο εργάζεται ως κολέγιο και επομένως είναι πολύ καλό ε, να προέρχονται ε, τα μέλη του από διαφορετικούς τομείς. Επίσης, ε, αν δει κανείς ε, την διαδικασία απαλλαγής, ε, αυτή τη στιγμή εργάζονται με τις qualified opinions. Πιστεύω ότι δεν θα πρέπει η πρόθεση της έκθεσης, της όποιας έκθεσης, να είναι μόνο τιμωρητική. Θα πρέπει να είναι και προληπτική αλλά και θεραπευτική να υποβάλλονται προτάσεις. Ε, δηλαδή βλέπεις ότι κάτι δεν λειτουργεί καλά, κάνεις ε, μία ε, έκθεση και λες ότι μπορεί στο μέλλον να αλλάξει αυτό και το άλλο και το άλλο και αν λοιπόν η κατάσταση βελτιωθεί στο μέλλον, αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Εγώ δεν πιστεύω ότι η έκθεση θα πρέπει να είναι name and shame ή έκανες εκείνο, έκανες το άλλο και θα τιμωρηθείς. Επομένως είναι καλό να ε, δουλεύει κανείς ε, σε ε, ένα υψηλό επίπεδο, σε ένα υψηλό επίπεδο. στις περισσότερες περιπτώσεις, το 50% των περιπτώσεων, έχουμε ελάχιστα τα οποία είναι κάτω από το 50% και μόνο στο υπόλοιπο 50% έχουμε λάθη πάνω από το 50% οι αστοχίες οι οποίες είναι πάνω από το 50%. Επομένως, ε, τα πράγματα πρέπει να μην είναι μόνο άσπρα ή μαύρα. Ε, η πραγματικότητα πολλές φορές έχει πολλές αποχρώσεις ανάμεσα από το μαύρο και από το άσπρο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπαλσίτης. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητή κυρία Bomb. Ε, δεν έχω καμία αμφιβολία για την εμπειρία σας προσωπικά όπως ε, και πολλοί συνάδελφοι χαιρόμαστε για το ότι θα βελτιωθεί η ισορροπία των φίλων. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Είχατε αρκετά μεγάλη εμπειρία σε διάφορους τομείς, όπως και άλλα μέλη του ελεγκτικού συνεδρίου αλλά επίσης ε, ήσασταν και υπουργό και μέλος ε, του οργανισμού Λιμένος Αμβέρσας και επίσης ε, του Δημοτικού Συμβουλίου της Αμβέρσας. Δεν θεωρείτε ότι υπάρχει εδώ πέρα κάποια σύγκρουση συμφερόντων. Η δεύτερη ερώτηση σχετίζεται με την πρώτη. για τις ε, πληροφορίες ε, υψηλής ποιότητας ε, και για τους ευρωβουλευτές και την Κομισιόν. Το ελεγκτικό συνέδριο, όπως υπόθηκε, δεν μπορεί να έχει σωστές γνωμοδοτήσεις γιατί αρκετά κράτη-μέλη δεν στέλνουν σωστές πληροφορίες. Εσείς έχετε κάποια εμπειρία Θεωρείται λοιπόν ότι πρέπει να έχουμε σαφείς ε, πληροφορίες στις περιπτώσεις όπου παρέχουμε τέτοιες ε, πληροφορίες θα πρέπει οι ελεγκτικές υπηρεσίες να λαμβάνουν και την άμεση ευθύνη για κάτι τέτοιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά πως ε, και γνωρίζετε ότι ε, αν γίνω μέλος του Ελεκτικού Συνεδρίου, θα παραιτηθώ από όλες μου τις ιδιότητες ούτως ή άλλως έφυγα από την βελγική κυβέρνηση πριν από δύο χρόνια. Οπότε δεν είναι ότι έρχομαι από αυτή την θέση κατευθείαν στο ελεγκτικό συνέδριο και ήμουν και μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών του Βελγικού Κοινοβουλίου και θα παρτιθώ όπως σας είπα και από το, Βελγικό, το Δημοτικό Συμβουλίο της Ανδέρσας και τον Οργανισμό Λιμένος και εντάξει, αν υπάρξει κάποια ειδική έκθεση για τις ε, θαλάσσιες μεταφορές που αφορά την Ανδέρσα προφανώς ε, θα αναλάβει κάποιος άλλος συνάδελφος ε, τον συγκεκριμένο έλεγχο για να μην υπάρχει οποιαδήποτε υπόνοια ε, σύγκρουση συμφέροντων. Αλλά, όπως σας είπα, θα παραιτηθώ ξεκάθαρα από όλες μου τις θέσεις. Γεγονό επίσης είναι ότι συχνά είναι δύσκολο να έχουμε περίπλοκες ε, πληροφορίες και κάποια φορά γίνονται ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα αν ε, θέλουμε π.χ. να δούμε το τι κάνουν τα κράτη-μέλη για την ανεργία στην χώρα τους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί σε κάποιες χώρες ε, το θέμα είναι η ανεργία των νέων, σε άλλες χώρες είναι η ανεργία των πιο ηλικιωμένων και έχουμε διαφορετικά δεδομένα που πρέπει να τα συνδυάσουμε και να γίνει μία ανάλυση εις ε, βάθος ε, τελείως διαφορετικών και περίπλοκων δεδομένων. Μια πιθανότητα λοιπόν θα μπορούσε να είναι να συνεργαστεί το ελεγκτικό συνέδριο στενότερα με τις εθνικές ελεγκτικές αρχές. Υπάρχει ήδη μια επιτροπή επαφής ε, όπου έχουμε πολλές συναντήσεις αλλά νομίζω ότι καλό θα ήταν και οι εθνικές ελεγκτικές αρχές να κάνουν περισσότερους έλεγχους ε, στα συγχρηματοδοτούμενα έργα που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις εθνικές και τοπικές περιφερειακές αρχές. Θεωρώ λοιπόν ότι μια τέτοια συνεργασία θα μπορούσε να έχει ε, ως αποτέλεσμα γρηγορότερες και καλύτερες πληροφορίες. Βεβαίως είναι διαφορετικά τα πράγματα γιατί ήμουν ε, υπουργό Οικονομικών στην ε, φλαμανδική κυβέρνηση και αν το Βελγικό Ελεγκτικό Συνέδριο ήθελε περισσότερες πληροφορίες έστελνε απλά ένα email. Βεβαίως πρόκειται για μια μικρή περιφέρεια στην ε, μεγάλη Ευρώπη και εκεί είναι ευκολότερο βεβαίω να δοθούν τα δεδομένα. Γιατί δεν υπάρχει και τόση ποικιλομορφία στα δεδομένα που λαμβάνει το ελεγκτικό συνέδριο. Ευχαριστώ κύριο Στάς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα μιλήσω Ολλανδικά και για να δουλέψουν λίγο διερμηνείς και για να ακούσει και η κυρία Τούρτελμπομ την γλώσσα της. Λοιπόν, Πριν έρθετε συζητήσαμε την απαλλαγή της Κομισιόν και η είναι ο κύριος Τσέλερ και κάποιες παρατηρήσεις που κάνει ο κύριος Τσέλερ είναι το γεγονός και η ανησυχία ότι η Κομισιόν όλο και περισσότερο εργάζεται με νέα χρηματοδοτικά μέσα, με ταμεία όπου τελικά η διαφάνεια και ο δημόσιος έλεγχος της χρήσης των κονδυλίων γίνεται προβληματικός και στην συνάντησή μας με τα μέλη του ελεγκτικού συνεδρίου πριν από λίγες εβδομάδες ε, συζητήσαμε με τον κύριο Ντένις Ντεγιόγκ της ΓΚΟΕ Είπαμε πως ε, το ελεγκτικό συνέδριο ε, έχει περιορισμένη πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Βλέπουμε λοιπόν μια τάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πως δημιουργούνται άλλα μέσα εκτός του προϋπολογισμού, διάφορα ταμεία, έχουμε την αυξανόμενη ισχύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπου δεν έχει ε, πολλές αρμοδιότητες στο ελεγκτικό συνέδριο, ούτε εμείς ως Ευρωπαϊκό Βούλιο, πώς το βλέπετε και πώς το κρίνετε ως ε, πρώην πολιτικός και ως ε, μέλος ε, προσεχώς του ελεκτικού συνεδρίου. Τι θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει. Ευχαριστώ. Πράγματι, αν δει κανείς τις παρατηρήσεις του ελεγκτικού συνεδρίου για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, για την ε, διαχείριση του προπολογισμού και την ε, χρηματοοικονομική διαχείριση υπάρχει η παρατήρηση ότι πράγματι υπάρχουν πληρωμές ε, οι οποίες γίνονται εγκαίρως και κανονικά αλλά ότι επίσης υπάρχει μικρή ευελιξία και αυτό μας ανησυχεί γιατί υπάρχουν εκρεμείς δεσμεύσεις οι οποίες βεβαίως θα πρέπει να υλοποιηθούν ε, σε βάθος χρόνου στο πλαίσιο του πι δέλτα Γιατί βεβαίως ακούμε ότι χρειαζόμαστε όλο και περισσότερα ευρωπαϊκά ταμεία, χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερα και διαφορετικά μέσα χρηματοδοτικά και ακριβώς έχουν πρόβλημα αποτελεσματικής διάθεσης των κονδυλίων τα κράτη-μέλη και το γνωρίζουμε αυτό και από την Αμβέρσα, όπου είναι δύσκολο ακριβώς να υλοποιήσουμε κάποια πράγματα και είναι και μια τάση την οποία βλέπουμε και στα κράτη-μέλη, ότι δουλεύουμε όλο και περισσότερο με διαφορά ταμεία. Εντάξει, αφενός αυτό είναι απαραίτητο αν θέλουμε να προσελκύσουμε ιδιωτικά κεφάλαια, ότι δηλαδή πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και κάποια συγκεκριμένα χρηματοδοτικά μέσα αλλά αυτό το οποίο έχει σημασία είναι να υπάρχει διαφάνεια, να έχουμε την δυνατότητα του ελέγχου. Για εμένα λοιπόν ε, που είμαι πολιτικός ε, και έχω εργαστεί πολιτικός ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά γνωρίζω ότι όταν θα πάω στο ελεγκτικό συνέδριο η δουλειά μου είναι να συνεργαστώ με μια ολόκληρη ομάδα ανθρώπων για να συνεργαστούμε, να κάνουμε έλεγχο και να συντάξουμε μετά αποτελεσματικές ελέγχεις. Δηλαδή να λέμε αν τα πράγματα είναι αποτελεσματικά, αν υπάρχει διαφάνεια, είναι λοιπόν και ένα μέσο της σύγχρονης διαχείρισης και της κρατικής, αλλά η φάνεια είναι το κρίσιμο. Είναι προβληματικό αν δεν ξέρει κανείς ποια ταμεία βρίσκονται σε ποιες χώρες ε, και ποιες είναι και οι μακροπρόθεσμες, τα μακροπρόθεσμα ανοίγματα τα οποία υπάρχουν, κάτι το οποίο καμιά φορά δημιουργεί δυσάρεστες εκπλήξεις. Και αν πάω στο ελεγκτικό συνέδριο, οπωσδήποτε στο κομμάτι των παρατηρήσεων, των ε, ετήσιων εκθέσεων οπωσδήποτε θα πούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει και διαφάνεια για να κρίνουμε σωστά το τι συμβαίνει με τα ταμεία. Είναι βασικός κανόνας επίσης στην συνθήκη ότι το ελεγκτικό συνέδριο στηρίζει το κοινοβούλιο στο ελεγκτικό του έργο και στον έλεγχο του Συμβουλίου Υπουργών και της Κομισιόν. Έβαλα και το δικό μου το όνομα στην ε, ημερήσια διάταξη. Μου φαίνεται πολύ καλή η υποψηφιότητά σας μου. Χρειαζόμαστε περισσότερη εμπειρία σε θέματα μετανάστευσης. Επισκεφτήκαμε την Ελλάδα την προηγούμενη εβδομάδα σε δύο καταβλισμούς και ευχαριστώ και τους αδέλφους που ήταν μαζί μας που επισκεφθήκαμε και είδαμε ότι τα χρήματα που πάνε για τους μετανάστες τα βλέπουμε μόνο όταν έχουν φύγει πια και δεν ενδιαφέρεται κανείς πού αξιοποιούνται τα χρήματα αυτά. Είναι χρήματα που πάνε για τους ε, ε, για το νερό, για το φαγητό, για την ε, ε, αποχέτευση χάνονται. Χάνονται, Ξαφανίζονται, δεν είναι ωραία έκφραση, αλλά πάντως έχουν φύγει τα χρήματα αυτά και δεν είναι δυνατόν να προσμετρηθεί το που χρησιμοποιήθηκαν γιατί δεν έχουμε αρκετά δεδομένα. Γι' αυτό το λόγο χαίρομαι που έχετε αυτή την εμπειρία και θα αναλάβετε αυτή την εξειδίκευση του ΣΥΠΗΝ στο ελεγκτικό συνέδριο, γιατί για τα θέματα αυτά δεν έχουμε φτάσει στο βαθμό που θα έπρεπε, στο επίπεδο που θα έπρεπε. Έχουμε προβλήματα κοινά σε όλα τα κράτη-μέλη, στη Γερμανία, στην Ελλάδα. Βεβαίω είναι πιο οξυμένα τα προβλήματα, αλλά και η Ιταλία έχει αντίστοιχα προβλήματα. Και πρέπει να συμβάλλουμε κι εμείς. Και γι' αυτό στηρίζομαι στη δική σας την εμπειρία. Μια ερώτηση που διατυπώνω πάντα σε κάθε υποψήφιο. Τι θα μπορέσετε εσείς να προσφέρετε και αν θα ζείτε στο Λουξεμβούργο. Παρακαλώ κυρία Γιάλα Σέντερ. Ναι, ε, πραγματικά χρειαζόμαστε πολύ εμπειρία, περισσότερη εμπειρία. Ε, και οπωσδήποτε θα πρέπει, θα πρέπει οπωσδήποτε λέω να ε, υπάρχει κάποια στήριξη όπως είπα και προηγουμένως ε, είχαμε προβλήματα ε, όσον αφορά ε, την, ε, όσον αφορά την ομάδα μου και αμοιβέ υπουργών και τα λοιπά, θα ήθελα να υπάρχει έτσι ένα cooling off period, γιατί ε, σίγουρα διαφορετικά θα έχουμε πολύ μεγάλα προβλήματα. Εγώ θα έλεγα λοιπόν ότι στα πλαίσια της εμπειρίας σας ε, έχετε μεγάλη εμπειρία, το ξέρουμε, και πολύ ενδιαφέρουσες ε, και σε σχέση με την δικαιοσύνη κλπ να έχουμε μια cooling period γι' αυτό. Βεβαίω στα πλαίσια του κολεγίου του ελεγκτικού συνεδρίου ε, ε, θα την χρησιμοποιήσετε την εμπειρία σας γιατί διαφορετικά θα υπάρχουν αντιδράσεις από την ομάδα. Άρα, αν κατάλαβα καλά, υπάρχει αυτή η περίοδος ε, cooling off που έχει γίνει δεκτή. Έτσι, αν σας κατάλαβα καλά. Παρακαλώ, για να απαντήσετε. Ο εισηγητής όμως μετά. Με συγχωρείτε και αυτός. Ή θέλετε μετά. Με συγχωρείτε κυρία Τουρτουργού. Κύριος Ταράντ. Όχι, ας ολοκληρωθεί αυτή η ανταλλαγή. Και μετά θα κάνω ένα τελικό σχόλιο, αν μου επιτρέπετε. Κυρία Τούρτελμπομ. Ε, ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας για το θέμα της μετανάστευσης. Παραμένει βέβαια πολύ περίπλοκο και όχι μόνο για τους αρμόδιους για τη χαράξη πολιτικής, αλλά και αν πρόκειται να διατεθούν κονδύλια και υποστήριξη στα κράτη-μέλη που έχουν μεγαλύτερη πίεση και πάλι, και το έχει παρατηρήσει το Ελεκτικό Συνέδριο, δεν υπάρχουν δομές αναφοράς, λογοδοσίας, αυτή τη στιγμή ακόμη, για τους πόρους, αλλά και γενικότερα για τους πόρους για την προσφυγική κρίση, αλλά και γενικότερα στη διαχείριση της, ε, του μεταναστευτικού. Δεν υπάρχουν εκθέσεις αρκετά αναλυτικέ. άρα χρειάζεται βελτίωση, το, λέμε και σε εκθέσεις, το λέει και το Λεπτικό Συνέδριο στι εκθέσεις του, με τρόπο διπλωματικό. Μεταξύ 2008 και 2009 ήμουν υπουργό Μετανάστευση στο Βέλγιο. Πριν να ξεσπάσει η προσφυγική κρίση, ήδη είχαμε σε επίπεδο ε, υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης να συζητούμε την προοπτική μιας κοινή μεταναστευτικής πολιτικής στην Ευρώπη και πώς θα μπορούσαμε να στηρίξουμε τις πιο ευάλωτες χώρες να αντιμετωπίσουν αυτή την κρίση. Αυτές που έχουν δηλαδή μεγαλύτερες πιέσεις να υποστούν. Και βεβαίως συμφωνώ μαζί σας, όντως, αυτή τη στιγμή και το βλέπουμε ε, στην έκθεση ότι δεν είναι ακόμη σαφή συγκεκριμένη η διαπίστωση αν γίνεται σωστή διαχείριση των κονδυλίων. Αφενός μένει διότι ο προϋπολογισμός από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για τη μετανάστευση και την, ε, τους συνοριακούς ελέγχους ενισχύεται, άρα όλο και μεγαλύτερη θα είναι και η πίεση για το ελεκτικό συνέδριο να τον επαληθεύει, να ελέγχει την αξιοποίηση των χρημάτων του Ευρωπαίου φορολογουμένου, γιατί θα πρέπει να δείξουμε ότι αντιμετωπίζουμε την μεταναστευτική κρίση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, χρησιμοποιώντας τα χρήματά του. Ταυτόχρονα δεν είναι δυνατόν πάντα, δεν είναι ευχερές πάντα να συλλέγουμε τα κατάλληλα και ε, σωστά δεδομένα για το πώς δαπανήθηκαν τα κονδύλια. Πάλι βέβαια είναι και ένα καινούριο καθήκον, μια νέα αρμοδιότητα και δουλειά που μπορεί να γίνει σε συνεργασία και με τις χώρες εταίρους, όχι μόνο με τα κράτη-μέλη. Άρα θα προχωρήσει και με χαρά βλέπω ότι στην, ε, στο ετήσιο πρόγραμμα του 2018 βλέπουμε πέντε εκθέσεις να αναγγέλλονται για τα θέματα της μετανάστευσης και της ασφάλειας και όσο περισσότερες εκθέσεις επιδόσεων συντάσσουμε και καλύτερη εμπειρία συλλέγουμε, τόσο καλύτεροι θα είμαστε φαντάζομαι στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ και τώρα για να ολοκληρώσει ο εισηγητή. Α, όχι, ένα λεπτό. Για το Λουξεμβούργο. Πού θα μένετε, πού θα μένετε. Ναι, ναι, όχι στο Λουξεμβούργο, στο Λουξεμβούργο. Δεν είμαι σε θέση να πηγαίνω έρχομαι κάθε μέρα μεταξύ Αμβέρσα και Λουξεμβούργου. Η δε πρωτεύουσα, η πόλη του Λουξεμβούργου είναι πολύ όμορφη. Σε διαμέρισμα σε ξενοδοχείο, λέει η Όχι, σκοπεύω να ε, νοικιάσω ή να αγοράσω ένα διαμέρισμα. Αλλά πάντα θα μένω εκεί full time. Είναι καλό να μπορεί κανείς να γυρνάει σπίτι του μετά από μια σκληρή μέρα δουλειά. Και είναι και ευχαριστή η πόλη. Καλώς ευχαριστώ και ο εισηγητή για να ολοκληρώσουμε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολύ σύντομα σχετικά με αυτό το θέμα του cooling off της περίοδου Κρίμα που είναι το Βέλγιο βασίλειο και όχι ε, δημοκρατία. Γιατί, αν είναι ε, είναι λογικό και προβλέπεται ε, να παίρνει ακόμα χρήματα κάποιος από το ελεγκτικό συνέδριο κατά τη διάρκεια του, της cooling period, αλλά να είναι και ε, πρόεδρος ε, στη χώρα του ή να κατέχει κάποιο αξίωμα. Αυτό δεν είναι τόσο σωστό όπως είπε και ο κύριος Φλάνναγκαν, σκέφτομαι και εγώ ότι ίσως θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερους επαγγελματίες auditors αργότερα, αλλά δεν είναι ε, τη σημερινή συζήτηση σε αυτό. Ε, είναι πολύ καλό που έχουμε έναν καλό υποψήφιο και στρέφομαι σε εσά κύριε Φλάναγκαν. Είμαι πεπισμένος ότι δεν είναι όλοι οι πολιτικοί κακοί και το λέω γιατί σας βλέπω και σας έχω απέναντί μου. Yeah. Thank ευχαριστώ και έτσι ολοκληρώνουμε την ακρόαση. Και τώρα πάμε και κλεισμένο των θηρών προκειμένου να κάνουμε την ψηφοφορία. Παρακαλούνται οι μία έχοντες εργασία μέσα στα επόμενα πέντε λεπτά να αποχωρήσουν από την αίθουσα. Τα πέντε λεπτά αυτά οι ομάδες μπορούν να τα αξιοποιήσουν για τις διαβουλεύσεις τους. Και σας ευχαριστώ κυρία Τούρτελμπο.